Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλή δουλειά. liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Λοιπόν, συνάδελφοι, σας καλωσορίζω θερμά στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Τουλάχιστον όμως ε, ακυρώσαμε την ε, αυριανή συνεδρίαση. Φαντάζομαι σας βολεύει όλου αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει βεβαίω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξη. Έγκριση αυτή. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Όχι. Επομένως εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση της 3 η Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν στα έγγραφά σας τα πρακτικά, υπάρχουν παρατηρήσεις που θέλετε να κάνετε, σχόλια για τα πρακτικά, όχι. Θα πρότεινα λοιπόν να θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αν έως το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης δεν έχουν υποβληθεί σχόλια ή παρατηρήσεις. Σημείο 3. Ανακοινώσεις Προέδρου. Σήμερα έχουμε διερμηνία στις εξή γλώσσε. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Και να σας υπενθυμίσω, όπως πάντοτε, ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Θέλω επίση να σας δώσω κάποιε πληροφορίε σχετικά με το, τη 12η έκδοση του βραβείου Lux. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει επίσημα στις 15 Οκτωβρίου. Από την ημέρα εκείνη θα ξεκινήσει και η ψηφοφορία. Μπορείτε αφού δείτε τις ταινίες να ψηφίσετε. Ε, και ο κωδικός για το Video On Demand καθώς και το πακέτο DVD ε, σε περιορισμό αριθμό αντιτύπων βεβαίως θα είναι διαθέσιμο για τα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Την προηγούμενη χρονιά δυστυχώς πρέπει να πω ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία ήταν περιορισμένος, να το πω ευγενικά. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα ως Επιτροπή, να μιλήσουμε για τις ταινίε αυτές, να τις δούμε καταρχάς. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να ψηφίσουμε για το βραβείο Λούξ. Γι' αυτό και σας καλώ όλους να γίνεται ενεργή αγγελιοφόρη του βραβείου Λουξ. Όχι μόνο εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και εδώ, εντός των γραμμών των Ευρωβουλευτών. Για την ε, ε, επιλογή των ε, ταινιών που έχει γίνει βρίσκεται κάποιες πληροφορίες στα εγγραφά σας. Από ό,τι ενημερώθηκα, πρόκειται για τρεις πολύ διαφορετικές μεν ταινίες, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες ταυτόχρονα και έχω πραγματικά μεγάλη αγωνία να δω ποιος στο τέλος θα ε, ε, βραβευτεί. Τις πληροφορίες δεν θα σας τις δώσω τώρα για τις ταινίε, υπάρχουν όλα στα έγγραφά σας. Τις ε, ταινίε αυτές μπορεί να τις, ε, θα τις προβάλλουμε 15 με 19 Οκτωβρίου και 5 με 9 Νοεμβρίου, δύο φορές την ημέρα, στην αίθουσα Γεχούντι Μενουίν, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν κάποιες ε, εξαιρέσεις, αν θέλετε όμως να παρακολουθήσετε τις ταινίες αυτές στην προβολή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Ε, οι μέρες του βραβείου Λουξ θα πραγματοποιηθούν ε, επίσης και φέτος θα γίνουν πάνω από 200 προβολές σε ολόκληρη την Ευρώπη για χιλιάδες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε βεβαίως την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ε, τις ταινίες αυτές σε περισσότερα από 20 φεστιβάλ και χώρους εκδηλώσεων. Στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου θα προβληθούν οι ταινίες αυτές σε 15 διαφορετικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόγραμμα αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στην ε, συνεργασία μας με το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Στόχος είναι να ενισχυθεί η προβολή του βραβείου ε, Λουξ, να διευρυνθεί το κοινό. Οι τρεις σκηνοθέτες θα προσκληθούν και στις Βρυξέλλες θα έρθουν εδώ στο Μποζάρ, στις Βρυξέλλες και στο Cinema Galleries και από εκεί, μετά την προβολή των ταινιών τους θα συμμετάσχουν σε διάφορες συζητήσεις που θα γίνουν επί των ταινιών τους μετά την προβολή τους. Οι εκδηλώσεις αυτές θα μεταδοθούν και live στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Άρτε. Η διαδικασία της ψηφοφορία είναι η γνωστή, αυτή που έχει ακολουθεί και τα, προηγούμενα χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ε, καλείστε όλοι να ε, υποβάλλετε την ψήφο σας από τις 15 ε, Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου στην ε, ιστοσελίδα του βραβείου Λουξ και η απονομή του βραβείου θα γίνει ω συνήθως στο Στρασβούργο την Τετάρτη στις 14 Νοεμβρίου στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ε, πριν από την τελετή θα γίνει και ένα σεμινάριο για δημοσιογράφους ε, θα συμμετάσχει η Εύελιν Γκέπχαρτ, η αντιπρόεδρος, ε, η οποία έχει προσκαλέσει και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τον Βιμ Βέντερς, για να μιλήσουμε για δικαιώματα αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κινηματογράφου, με συγχωρείτε. Ελπίζουμε να επιβεβαιώσει και την παρουσία του ο Βιμ Βέντερς, είστε όλοι θερμότατα προσκεκλημένοι. Ε, να σας ε, υπενθυμίσω ότι πρέπει να υποβάλλετε έτοιμα αν θέλετε κωδικό για, τη διαδικασία, για την υπηρεσία Video On Demand για τις τρεις ταινίες για να τις δείτε διαδικτυακά. Είναι λίγο περίπλοκη αυτή η διαδικασία, δυστυχώς όμως είναι απαραίτητη διότι οι ταινίες αυτές βρίσκονται σε ένα σερβερ, σε έναν διακομιστή ο οποίος δεν βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά έχει ανατεθεί σε εξωτερικό πάροχο ε, υπηρεσιών η υπηρεσία αυτή Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο περίπλοκη, αλλά εφικτή η διαδικασία αυτή. Θα το ξαναδούμε βεβαίω και με τι υπηρεσίε μα, αν μπορούμε να επιστρέψουμε στην παλιότερη, στο παλιότερο καθεστώ, για να ε, μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε ευρωβουλευτή, χωρί να χρειάζεται να περνάει από αυτή τη διαδικασία υποβολή αιτήματο για κωδικό όχι μόνο για τη δική μας Επιτροπή, για όλους τους ευρωβουλευτές φυσικά. Δυστυχώ, όμως φέτος δεν κατέστη δυνατό να επιτύχουμε μια καλύτερη λύση. Να ευχαριστήσω τη Μαρισέλα και τον Γένριχ που ε, συνοδεύουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διαδικασία της απονομής ε, του ε, βραβείου Λουξ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, περνάμε επόμενη, στο επόμενο σημείο της ημερής σας διάταξης. Σήμερα έχουμε ψηφοφορία για πέντε νομοθετικές νομοδοτήσεις. Κυρία Λιμπάτσκα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα για το βραβείο Λούξ. Πέρσι είχα παραπονεθεί για, τις, για την ποιότητα των βίντεο κασετών μου είπαν ότι θα τα, μάλλον όχι την ποιότητα, για την ποσότητα που δεν λάβαμε εμείς. Είχαν, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα λάβουμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού. Also die Videos für die Abgeordneten soll es geben, äh, wohl... Ναι, θα υπάρχουν βίντεο για τους ευρωβουλευτές από τις 15 Οκτωβρίου και έπειτα, όπως είπα. Παρασκευή είναι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα ναι, εντάξει. Σα διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα για να περάσει η διαδικασία αυτή ομαλά, να λάβετε όλοι τα DVD και θα εξασφαλίσουμε βεβαίως τουλάχιστον τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού να λάβουν τα DVD. Ωραία, μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στις ψηφοφορίες τώρα. Όπως είπα, πέντε νομοθετικές γνωμοδοτήσεις έχουμε. Περνάμε κατευθείαν Ενδιάμεση έκθεση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27, η θέση του Κοινοβουλίου Ενόψη Συμφωνία. Εγώ ήμουν η συντάκτρια τη γνωμοδότηση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει για άλλη μια φορά. Του ε, συνεργάτε, του βοηθού ε, των πολιτικών ομάδων, ε, τη γραμματεία. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και καταλήξαμε σε ένα πολύ καλό κείμενο, θεωρώ. Και ελπίζω βεβαίως ότι ε, η ε, γνωμοδότηση αυτή θα ληφθεί υπόψη και από την Επιτροπή Προπολογισμού και στη συνέχεια συνολικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην ε, ε τροπολογία 1. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 4 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Θα περιμένω, θα περιμένω, ναι, μην ανησυχείτε. Ich wollte noch gefragt haben, ob alle ihr Kärtchen Ήθελα και να ρωτήσω και το ξέχασα αν έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί σας. So, die Abstimmung... ψηφοφορίας. Πέρας. 25 υπέρ, 4 αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση του Bogdan Venta, γνωμοδότηση με συγχωρείτε, για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη και ε, περνάμε με την τροπολογία 8. Με συγχωρείς πρώτα Μπόγκταν αν επιθυμείς να πεις κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, ιδιαίτερε ευχαριστίε στου χιώδη ηγητέ για την πολύ καλή συνεργασία για το θέμα μα. Πολλέ ευχαριστίε επίση για την βοήθεια για τη γνωμοδότηση στις ε, της Γραμματείας και βεβαίως και στην δική μου ε, προσωπική βοήθεια. Σας ευχαριστώ Μπόγκταν. Αρχίζουμε. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές ας υπαλληθεύσουμε το αποτέλεσμα 114 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος το Λαϊκό Κόμμα έχει μία πλεονάζουσα ψήφο. Κάποιος δηλαδή πρέπει να αφαιρέσει την κάρτα ψηφοφορίας εκ των μελών του Λαϊκού Κόμματος. Ωραία, τώρα είναι σωστή η αριθμή. Πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας απορρίπτεται ψήφι 15 κατά 13 υπέρ. 9 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας το επαληθεύσουμε ξαναλέω λοιπόν 117 πέρας. Απερίφθη λοιπόν πράγματι με την ίδια πλειοψηφία όπως πριν. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας επαληθεύσουμε Έναρξη της ψηφοφορίας. Τέλος. Απερίφθη 15 κατά 14 υπέρ. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας επαληθεύσουμε 146 έναρξη της ε, ψηφοφορίας <clears throat> τέλος όντως 14 υπέρ 10 κατά 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πηγαίνουμε στην 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 τώρα, 18. Και 150 γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 19 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 και 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 154 154 λοιπόν, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Αν με συγχωρείτε, απορρίπτεται η προηγούμενη, λέει ο Πρόεδρος. 155 τώρα, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά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 εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά σε παληθεύσουμε 171 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος 13 υπέρ, 15 κατά. 5 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές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 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πρόεδρος, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ,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 αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας το επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απερίφθη όντως 13 υπέρ 16 κατά 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ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 αποχές εγκρίνεται τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Όντως 12 υπέρ 16 κατά. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση αρχίζει 81 λοιπόν. Τέλο ε, συγγνώμη, 17 υπέρ, 12 κατά. Συγγνώμη, δεν είχα ε, πλήρη εικόνα. Τώρα, 82 υπέρ, κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι απόλυτα βεβαία ας αρχίσουμε λοιπόν την επαλήθευση τέλος 15 κατά, 14 υπέρ, απερίφθη. 95 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά. Αποχές, παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια, καθαρά τα χέρια, για να μπορώ να βλέπω την εικόνα πλήρω. Δεν έχει πει η πρόεδρο γιατί ανοίγει την ψηφοφορία, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει κάνει. Έχετε αποκοιμηθεί όλοι, ρωτάει η πρόεδρο. Τέλο τη ψηφοφορία. Ισοψηφία 14-14 απορρίπτεται. 100 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ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 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλίση αρχίζει Τέλος, 27 ψήφοι υπέρ, μία αποχή και καμία ψήφους κατά. Συγχαρητήρια, Μπόγκταν. Και ακολουθεί η έκθεση Λουίτζι Morgano. Για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Λουίτζι, θέλεις να τοποθετηθείς, να πεις κάτι. Παρακαλώ. Sì, molto brevemente, davvero un sentito ringraziamento. Εντάχει θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες και ιδιαίτερα τους κοιόδης για τη συνεργασία του, στη γραμματεία ιδιαίτερα. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική και έτσι φτάσαμε σε μία συγκεκριμένη πρόταση από την δική μας Επιτροπή. Ευχαριστώ. Äh, Luigi Ευχαριστούμε, Λουίτζι, για το έργο σου και περνάμε με, στην τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε αυτό ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά επί τη 86 πέρας απορρίπτεται με 15 ψήφου, κατά 3 υπέρ 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Ε, απεσύρθη. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. αποχέ. καλύτερα να τα δούμε ηλεκτρονικά αυτό. Ψηφίστε παρακαλώ με τι καρτούλε σα. Geschlossen. Mit 15 Απορρίπτεται. 15 κατά, 13 υπέρ. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές ε, ψηφίζουμε ξανά για την 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ ξέχασα κάτι 103. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108. Υπέρ, κατά,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 αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε αυτό επαληθεύουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ geschlossen πέρας απορρίπτεται 16 κατά 11 υπέρ 129 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Ψηφίσουμε τι τις τροπολογίες 133. 133. Ξαναλέω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές ξανά υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά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 Συμβιβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Κανένα πρόβλημα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, 13 κατά. Συμβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61. Υπέρ, κατά αποχές που καλύτερα να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά δεν είμαι βέβαιη ψηφίζουμε παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7, 67 ε, με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 75. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά αποχές καλύτερα να το ελέγξουμε αυτό ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 80 παρακαλώ ψηφίστε πέρας ψηφοφορίας 14 υπέρ 14 κατά απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση ηλεκτρονικά ψηφίζετε παρακαλώ για το σύνολο της γνωμοδότησης. Geschlossen. Mit 28 ja. Πέρας. Υπέρ 28, μία αποχή εγκρίνεται. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια. Dann kommen wir jetzt zum, zur Stellungnahme zum Europäischen Regionalfonds. Berichterstatterin war Marlene Mitzi. Marlene, möchtest du, möchtest du noch Αχ, δεν είχα. Εντάχει θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες ε, για αυτό το θέμα και ιδιαίτερα τους σκιώδεις. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα έγγραφο που είναι πολύ σημαντικό για τις περιφέρειες και υπο, τις υποστηρίζουμε βεβαίως στεναρά. Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρλέν. Ψηφίζουμε επί τη ε, γνωμοδότηση για τι ειδικέ διατάξει για το στόχο τη Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία με τη στήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη. Νομίζω ότι είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα πριν, γι' αυτό το ξαναλέω. Wir Τροπολογία 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42. Υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά,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 αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά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 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 147 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 148 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 152 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 153 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 154 υπέρ κατά αποχές απόρριψη. Επίσης 132 υπέρ κατά αποχές απόρριψη. 22 υπέρ κατά αποχές απόρριψη. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία δωρεάν μασάζ για τη γλώσσα μου. Ήταν όλο αυτό, λέει η πρόεδρο. Τέλος τη ψηφοφορία. Ψήφι 23 υπέρ, 3 αποχέ και μία ψήφο κατά. Με μεγάλη λοιπόν πλειοψηφία εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Και ακολουθεί η τελευταία ψηφοφορία που και αυτή είναι μακροσκελεστάτη. Θα προσπαθήσω να προχωρήσω με την ίδια ταχύτητα και μιλούμε για την γνωμοδότηση για την προστασία προσώπων που καταγγέλουν παραβιάσεις ενωσιακού νόμου. Η συγητής είναι ο κύριος Μαλτέζε που δυστυχώς κολλείεται σήμερα διότι ασθενεί. Του ευχόμαστε περαστικά και νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην την ψηφοφορία με τη συμβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.14 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 264 θα ψηφίσουμε. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε επί τη τροπολογία 78. Υπέρ. Απερίφθη και γι' αυτό δεν καταπίπτει η 78. Και ψηφίζουμε επί της, τρο... Ε, τροπολογίας 78. Υπέρ. Απερίφθη, λέει η Πρόεδρος. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2,70 υπέρ, κατά... Α, όχι, όχι, δεν ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 2,70. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22. <laughs> wollte sagen, ihr habt doch richtig geguckt. Also, Kompromiss 21. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 299. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Achso, Entschuldigung, den habe ich übersehen. Entschuldigung, es ist viel, den habe ich übersehen. 300, äh, dafür. 300, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην συμβαστική 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 312. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 3.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.17 υπέρ κατά αποχές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 εγκρίνεται. 3.24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. 3.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Επιστροπολογίες 5. Schon ganz durcheinander. Geschlossen. Πέρας. Εγκρίνεται. 14, 13 κατά. Και περνάμε στη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ, κατά, άμα δεν σηκώνετε τα χεράκια σας, δεν μπορώ να βλέπω τι ψηφίζετε. Υπέρ τις 10. Τροπολογία 10. Υπέρ. Ένα. Geschlossen. τη Εγκρίνεται 18 υπέρ 9 κατά. Δεν το έβλεπα όμως γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σας καθαρά για να βλέπω. Λοιπόν, 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 126 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να το επαληθεύσουμε αυτό ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 126 ψηφίστε παρακαλώ τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 υπέρ 14 κατά 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ ε, και 129 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130 και 131 μαζί υπέρ, κατά, αποχές Καλύτερα να το επαληθεύσουμε αυτό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Geschlossen. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ, 13 κατά. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Βλέπω να κουράζεστε. Ας το ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Geschlossen. Mit 15 zu 11 angenommen. Εγκρίνεται 15 υπέρ 11 κατά. 136 dafür. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 21 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Dann prüfen wir das. Ας το ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Mit 14 zu 13. Εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ όχι συγγνώμη 28 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να το ελέγξουμε αυτό. Πέρας της προφορίας. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 13 κατά. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Geschlossen. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 12 υπέρ, 14 κατά. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ωραία, ας το ελέγξουμε λοιπόν, αφού υπάρχει διαφωνία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Geschlossen. Πέρας. Εγκρίνεται 17 υπέρ 10 κατά. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε. Πέρας, συγγνώμη, μεγάλη διαφορά, 22 υπέρ, μία ψήφο κατά, εγκρίνεται. Ist dann ein Problem. 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί του συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης. Πέρας τη ψηφοφορίας εγκρίνεται 24 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον συντάκτη της γνωμοδότησης αυτής. Ωραία. So, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit aufholen, wird mir gerade gesagt. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα. Με ενημερώνουν. Okay. Dann machen wir jetzt ganz schnell, weil... Πάμε γρήγορα. Γιατί η Σιλβί Γκυγιόμ πρέπει να τρέξει να πάει στη Λίμπε, γιατί και εκεί θα συζητήσουν το θέμα αυτό. Είμαστε στο σημείο 9 Τη σημερινές διάταξη. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ να το κάνετε ησύχω. Λοιπόν, σχέδιο γνωμοδότησης για το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Δικαιώματα και αξίες», Ταμείο Values. Συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η Σιλβί Γκυγιόμ, στην οποία και θέλω να δώσω το λόγο. Συγγνώμη, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε. 18. 18 Οκτωβρίου, 2 το μεσημέρι, είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Εμεί έχουμε ε, αποκλειστικά δικαιώματα για το δικό μας, για το παλιό πρόγραμμα «Η Ευρώπη των Πολιτών». Σίλβι Κιγιόμ, έχει το λόγο για να μας ε, παρουσιάσει τι προτάσει σου για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ Πέτρα. Ε, πρέπει να πάω στη Λίμπε, αλλά και εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε επί 20 λεπτά για την έκθεση Μποντίλ Βαλέρο, γι' αυτό θα είμαι κάπως τηλεγραφική. Ε, εδώ και καιρό ανταλλάξαμε απόψεις, ε, συντάχθηκε και γνωμοδότηση σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες που ε, συνεργάστηκαν υποπίεση και δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε διαβουλεύσεις ή ακροάσεις. Αυτό θα ήταν υπέρ ε, της κοινωνίας των πολιτών. Λυπούμαστε γι' αυτό. Τηλεγραφικά λοιπόν για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Για να πω καταρχήν ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση του παλαιού προγράμματος Ευρώπη των Πολιτών. Γιατί ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία για να προωθήσουμε την ε, συμμετοχή των πολιτών και για να ενισχύσουμε και το δημοκρατικό αίσθημα των πολιτών. Είναι ένα σημαντικός φάκελος επί του θέματος. Το δεύτερο, που αποτελεί συνέχεια του πρώτου, δεν είναι αποκλειστικά συμβολικό. Θα ήθελα να επανεισαγάγουμε στον τίτλο αυτή την έννοια της ηθαγένειας που δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή η ηθαγένεια, δικαιώματα και αξίες. Αυτός θα είναι ο τίτλος, ενώ τώρα μιλάμε για δέσμευση μόνο και συμμετοχή των πολιτών. Δεν είναι συμβολικό λοιπόν, είναι ουσιαστικό. Ως προς τον προϋπολογισμό θα πρέπει να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του για να είμαστε στο ύψος του ε, διακυβεύματος. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια ευρώ καταρχήν που έχουν εγγραφεί που αντικατοπτρίζει την κατάσταση. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς του προϋπολογισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μέρος των χρημάτων για πολιτική επικοινωνίας. Το τέταρτο σημείο για τον ορισμό των προτεραιοτήτων έχει ως εξής. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, συμμετάσχει σωστά ε, σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό θα ήθελα οι εκτελεστικές ε, πράξεις να αντικατασταθούν από κατεξουσιοδότηση πράξης. Επίσης, τις τροπολογίες δεν θα πρέπει να προβούμε σε ένα συναγωνισμό σε σχέση με τα μέτρα που αφορούν τις μεγάλες ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να ισχύσει για τις μικρές ε, εδαφικές οντότητες για να λειτουργήσει καλά αυτό το πρόγραμμα. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την εκτέλεση του προγράμματος σε αυτό τον ενδυνάμει ανταγωνισμό και θα πρέπει να δούμε και την προσβασιμότητα στο πρόγραμμα από ΑΜΕΑ τις τρίτες χώρες που συμμετέχουν επίσης ε, σε ενδεχόμενα προγράμματα και να μας απασχολήσουν ε, και τα σημεία επαφής των ε, εθνικών αρχών. Αυτά είναι τα έξι σημεία που θα ήθελα να θίξω καταρχήν και θα ήθελα να τελειώσω με ένα τεχνικό καθαρά ζήτημα. Ως προς το δημοσιονομικό δελτίο της Κομισιόν για την κατανομή δηλαδή των κονδυλίων. Μιλάμε για τις δεσμεύσεις και συμμετοχή των πολιτών καθώς και της ΜΚΟ που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση ΖΙΣΤ που εκπροσωπεί το 20% των οργανώσεων. Για ποιες οργανώσεις πρόκειται. Πρόκειται για το παλαιό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Just για την ισότητα των δύο φύλων και για τις ίδιες ευκαιρίες. Θα θέλαμε λοιπόν να είμαστε σίγουροι για τη συμμετοχή των πολιτών και πιστεύω ότι υπάρχει ένας επιμερισμός που δεν είναι απόλυτα σαφής. Θα ακούσω φυσικά την άποψη των σκιωδών για να ενισχύσω αυτό το πρόγραμμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Αυτά, Πέτρα. Ευχαριστούμε Σιλβί. Περνάμε τώρα στους οι εισηγητές. Ξεκινάμε με τον κύριο Μαλίνοφ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας παρακαλώ μην τα ξεπεράσετε όμως. Ναι, καταλαβαίνω. Θα ήθελα να αρχίσω με το θέμα του τέλους παρουσίασης της κυρίας Γκυγιώμα. Χτες συναντηθήκαμε με ΜΚΟ μετά από οργάνωση εκδήλωσης από τον κύριο ε, Μπόνι και την ε, Μποντίλ Βαλέρο των Πρασίνων. Θέλουμε να επικεντρωθούμε για να έχουμε του, τα κονδύλια σε ένα σημείο. Η ΜΚΟ μας παρουσίασαν υπολογισμούς αναφέροντας ότι τα χρήματα τελικά θα είναι λιγότερα. Η Επιτροπή είπε ότι υπάρχει κατακαιρματισμός και περιορισμένοι πόροι και γι' αυτό θα ήθελα να προσθεθούν περισσότερα χρήματα σε όλα αυτά τα προγράμματα. Αυτός είναι ένας από τους κινδύνους που υπάρχουν Και προσωπικά θα ήθελα να πω από οργανώσεις νεολαίας ότι το όλο θέμα μπορεί να συνδεθεί με το Erasmus Plus γιατί πρόκειται για αξίες, εκπαίδευση και κατάρτιση για καλύτερη συνέργεια. Και το τρίτο θέμα, επειδή βιάζομαι, είναι ότι υποστηρίζω τις τοπικές μικιο Επιμένω λοιπόν ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτές. Υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού, προαναφέρθηκε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι οργανώσεις των πολιτών θα πρέπει να είναι στο προσκήνιο. Δεν υπερεύει τα δύο λεπτά. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαρή Τερέζ. Έχουμε στόχο να προωθήσουμε το διάλογο μεταξύ Ευρωπαίων μέσα στα πλαίσια μιας αμεβαίας κατανόησης, στα πλαίσια της υπάρχουσας ε, δυστυχώς μυσαλλοδοξίας. Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση σε ευρωπαϊκά θέματα, άρα μας απασχολούν ε, τα θέματα αυτά εν ώψη των ε, μελλοντικών ευρωεκλογών θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα. Να δούμε ιστορικά, το ιστορικό μάλλον αυτών των προγραμμάτων μέσα στα πλαίσια της καλύτερης κατανόησης του παρόντος να δούμε και το θέμα της ε, δημοκρατικής ηθαγένειας και την κοινωνία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για να υποστηρίξουμε τις ανοιχτές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Μιλάμε, Μαρή Τερές, μπορείς να μιλάς πιο αργά, σε παρακαλούμε, αν θέλεις να σε παρακολουθούμε. Ε, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες. Ο συνάδελφος Μαλινόφ έκανε πολύ συνετές προτάσεις. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια ε, Σιλβί γιατί η έννοια της ηθαγένειας δεν υπάρχει πια στον τίτλο. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τους πολίτες. Γι' αυτό η λέξη ηθαγένεια θα πρέπει να επανεισαχθεί στον τίτλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ Πέτρα και ευχαριστούμε την εισηγήτρια βιάζεται και θα είμαι σύντομη. Το θέμα αυτό είναι ζωτικής ε, σημασίας για τις επικείμενες εκλογές και το κράτος δικαίου που είναι η πολιτική βάση των δράσεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις γειτονικές χώρες. Πρόκειται για την ενίσχυση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των μειονοτήτων ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Θέλουμε λοιπόν οι μειονότητες να μπορέσουν να αυτοενισχυθούν και να μην ε, υπάρχει, να μην υποστηριχθεί ο υφέρπον και αναδιόμενος εθνικισμός, γιατί αυτό στο τέλος σημαίνει πόλεμο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει στον τίτλο να, στον τίτλο να εμπεριέχεται η λέξη πολίτες, θα πρέπει να τονιστεί και θα μπω στις λεπτομέρειες των τροπολογιών μου για ε, τον προϋπολογισμό, μιλάμε για το πολιετές, υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη με το Συμβούλιο, αλλά υπάρχει συνδεσιμότητα και τα προγράμματά μας ε, είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν τα κονδύλια, κάτι το οποίο θα, θα αναφερθεί και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστούμε Χέλγα. Η κυρία Μπίλντ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση, κυρία Γκυγιόμ. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με και με τις ε, υποσύνδεση χώρες. Θεωρώ ότι η Ευρώπη ε, για τους πολίτες αποτελεί μία φιλοευρωπαϊστική προπαγάνδα. Αυτό γίνεται και με την αδελφοποίηση πόλεων. Μιλάμε για στερεότυπα μειονοτήτων και μεταναστών στη Σικελία. Υπάρχει ευρωσκεπτικισμός και δυστυχώς βλέπουμε μία αναζωπήρηση των ε, εθνικισμών και στη Σερβία. Η μάχη του Βερντέν έχει απορριφθεί. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι καταβλισμοί των μεταναστών. Η Ουγγαρία και η Πολανία είχαν μεγάλες αιτήσει. Η Ουγγαρία συνέλεξε το 17%. Πρόκειται όμως για εθνικό παρεμβατισμό και δεν δέχομαι κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. So, ε, ε, Entschuldigung, Silvia, bitte versuch's mal in Minute. Ναι, σε ένα λεπτό μόνο, Σίλβια. Ναι, ναι, ναι, εντάχει, εντάχει. Για τη Σίλβη θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι αυτά που προείπε εκτιμώ το σχέδιο που αναφέρεται στα σημαντικότερα σημεία. Μας ενδιαφέρουν ε, τα κονδύλια τα οποία ακολουθούν φθήνουσα πορεία. Η διαχείριση θα πρέπει να είναι καλύτερη. Δεν μπορεί να όλα, όλα να βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Just. Δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από εκείνη το πρόγραμμα. Θα πρέπει να εισαχθεί ο όρος ηθαγένεια στον τίτλο και θα πρέπει να ξέρουμε για ποιες οργανώσεις πρόκειται. Για διαφορετικά οι πολίτες δεν θα ξέρουν σε ποιον απευθύνονται. Και ένα ερώτημα. Ωραία η προσέγγιση bottom-up, Δεν κατάλαβα όμως κατά πόσο η πρόταση της Σιλβιή Γκυγιόμ είναι να μην ανοίξουμε το πρόγραμμα προς τρίτες χώρες. Ξέρω ότι αυτό ίσως είναι μία εμονή, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει συμμετοχή ή όχι. Ωραία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σιγκάν, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει κυρίως στο βασικό ερώτημα. Από πού προήλθε αυτό το 20%? Πώς αιτιολογείται? Για ποιο λόγο επελέγει μια τέτοια περίπλοκη διαχείριση των χρημάτων και γιατί δεν είχε ξεκαθαριστεί αυτό εξ αρχής, ε, στο κείμενο μέσα και επελέγει να ε, κρυφτεί το όλο θέμα κάπου σε κάποιο παράρτημα. Ενδεχομένως ε, με σκοπό να μην το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιος είναι ο λόγος, ποιο είναι το σκεπτικό αυτού του πολύ περίπλοκου μηχανισμού διαχείρισης των χρημάτων. Ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας στη συζήτηση για το, για το πρόγραμμα Ευρώπη, ε, των Πολιτών. Βεβαίω το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται μέχρι το 2020, άρα σημαίνει αυτό ότι έχουμε άλλα δύο ετήσια προγράμματα, το 2019 και το 2020. Και βεβαίως την περίοδο αυτή ε, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά, θα συνεχίζει να εφαρμόζεται, ε, θα χρησιμοποιήσουμε βεβαίως και το εργαλείο της ενδιάμεσης αναθεώρησης για να το βελτιώσουμε. Είναι δύο χρόνια, δεν είναι καθόλου μικρό το χρονικό διάστημα και μάλιστα είναι τα δύο χρόνια μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναγνώριση της σημασίας αυτού του προγράμματος και την ε, αναγνώριση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει σε αυτόν τον καιρό πριν από τις ε, ευρωεκλογέ και έχουμε σημειώσει όλες τι ε, τις παρατηρήσεις σας, τις συζητήσεις που έχουν, που έχουν γίνει για τις προτάσεις μας που ξέρετε ότι σκοπός ήταν να ε, διαρθρώσουμε το μελλοντικό σύστημα με έναν ορθολογικό τρόπο και να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις συνέργειες. Αυτό εξηγεί και τον ευσύνοπτο χαρακτήρα του κειμένου σχετικά με τα ονόματα, τις, ε, και, τις, και τους ε, σχετικά περιορισμένους ορισμούς που χρησιμοποιούμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά που έχετε κάνει, τις παρατηρήσεις σας, για το πρόγραμμα, για την εφαρμογή του. Ήταν ε, ένα απτό παράδειγμα και αποτέλεσμα καρπός της συνεργασίας μας τα τελευταία χρόνια. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις τροπολογίες που έχετε υποβάλει για τη βελτίωση του κειμένου, για τον προϋπολογισμό και το ύψος του. Κάθε ε, πρόγραμμα βεβαίως ε, θα ήταν ε, ικανοποιημένο αν είχε περισσότερα χρήματα στη διάθεσή του. Η Κομισιόν προτείνει αυτό που εκτιμήθηκε ότι θα ήταν διαθέσιμο, συνυπολογίζοντας και συνεκτιμώντας γενικά τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κομισιόν. Για τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία, μία από τις ιδέες για το νέο πρόγραμμα ήταν να αξιοποιηθούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων και ε, διαστάσεων των προγραμμάτων και νομίζω ότι θα φανεί στην πράξη, στη ζωή, ε, αν ήταν καλή η πρότασή μας αυτή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ενημερώσουμε όλους τους δικαιώχους για την ύπαρξη αυτού του προγράμματος για να το αξιοποιήσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ο τρόπος που βρήκαμε για να απαντήσουμε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη των, ε, της κοινωνίας των πολιτών. Αντί λοιπόν να ε, επιλέξουμε ένα μείγμα δικαιούχων μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιλέξαμε να ε, δώσουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα μπορούσε να αποφέρει αποτελέσματα σε όλους τους δικαιούχους. Το 20% ε, προτείνουμε να ε, υποβληθεί σε διαχείριση εσωτερικά στην Κομισιόν για να κατευθυνθεί ε, στη συνέχεια σε διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις <laughs> στη βάση των κριτηρίων. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο. Να σας πω και για την διεθνή συνεργασία με τρίτες χώρες και το γεγονός ότι τώρα στην τρέχουσα πρόταση πράγματι κάποιοι από τους εταίρους μας δεν υπάρχουν πλέον. Μιλώ για τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων για παράδειγμα. Θέλω να σα υπεβεβαιώσω ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση που έγινε ε, αξιολογήθηκε θετικά η συνεργασία αυτή και προκειμένου να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα χρειάζεται να υπάρχουν πάντοτε οντότητε φορεί και ε, στην, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνεργάζονται με του εταίρους μα στα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστεί η πραγματική αξία ε, αυτή τη συνεργασία. Και τέλος θέλω να πω ότι θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ξέρετε ότι ε, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να προσερχόμαστε εδώ στην Επιτροπή και να συναντιόμαστε με ευρωβουλευτέ για να δίνουμε εξηγήσει, να απαντάμε και να διευκρινίζουμε ζητήματα που σχετίζονται με τις προτάσεις μας. Όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σα. Και βεβαίω να ευχηθούμε κι εμεί ότι καλύτερο για το πρόγραμμα στο μέλλον. Η Ευχαριστώ πολύ για τι εξηγήσει σα. Θα χαρούμε ιδιαίτερω εφόσον δούμε ότι καταβάλει προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη μα, υπόψη τη, συγγνώμη, τα ψηφίσματά μα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναμένουμε περισσότερη υποστήριξη για τι μη κρατικέ οργανώσει. Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί εξήγηση για ποιο λόγο το 1 πέμπτο των κονδυλίων που θα έπρεπε να πάνε στο Citizens Program αποδεσμεύονται και τα διαχειρίζεται άλλη γενική διεύθυνση. Από τη δική μου σκοπιά αυτό σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό και το αντίθετο από μια προσπάθεια δημιουργίας συνεργειών και περιπλέκει το όλον διότι χρειάζεται εκ νέου συντονισμός μέσα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προφανές για μένα και νομίζω δεν είναι προφανές ούτε και για τις και τους συναδέλφους εάν ε, ρίξω μια ματιά στα πρόσωπά τους να πω τώρα και μια φράση για αυτή τη μαγική ορολογία. Συνέργειες και συμπληρωματικότητες, είπε η Επιτροπή. Ωραία ακούγονται όλα αυτά. Συνέργειες και συμπληρωματικότητες, αλλά μήπως μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει πώς φαντάζεται ότι θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Έχω στείλει και επιστολή στον Επίτροπο Έτιγκερ ήδη από τον Ιούνιο, έκτο Ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση, διότι προφανώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδής γνωρίζει τι πάει να πει οι συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ των προγραμμάτων. Και αν ε, τελικώς εγκρίνουμε κάτι τέτοιο, θα θέλουμε πριν να το κάνουμε αυτό να γνωρίζουμε εάν όντως δίνουμε λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να μετακινεί κονδύλια από εδώ και από εκεί. Κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Διότι εν τέλει εμείς θεσπίζουμε τις πολιτικές προτεραιότητες στη συνεργασία με το Συμβούλιο Υπουργών. Αυτή λοιπόν η έννοια συνέργειας και συμπληρωματικότητες, αυτές οι έννοιες, μήπως είναι απλώς κενά και λήφη λέξεων όπου πίσω δεν κρύβεται τίποτε άλλο παρά να δοθεί μια ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χειρίζεται τα κονδύλια όπως αυτή επιθυμεί. Η Σαμπίνε Φερχάιν. Γι' αυτό που είπες, συνέργειες και συμπληρωματικότητες. Δεν πρόκειται για τίποτε το νέο. Τα είχαμε και στα προηγούμενα προγράμματα, τα οποία κινούνται ακόμα. Είχαμε πει ότι βεβαίω και πρέπει να συμπληρώνονται τα προγράμματα μεταξύ τους σε ό,τι αφορά του στόχου, και ούτε επιτρέπεται το ένα πρόγραμμα να υπονομεύει το άλλο ω προ του στόχους. Όπω όπως, είπες, όπως όμως είπες και εσύ, εάν η ευελιξία αυτή σημαίνει μετακίνηση κονδυλίων δόθε κήθε, αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε. Όχι λοιπόν λευκή επιταγή. Συνέργειες ναι, συμπληρωματικό χαρακτήρα των προγραμμάτων, ναι, αλλά με συγκεκριμένο στόχο. Και ότι ζητείτε από τις χώρε μέλη να πάρουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα και τις στοχεύσεις τους και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ομογενοποιήσουν, αυτό νομίζω για μένα είναι απολύτω αυτονόητο. Ευχαριστώ. Σίλβι Γκυλιόμ. Για να απαντήσω σε, στις υποψήφιες χώρες, Συμφωνώ ότι οι χώρες αυτές δεν αποκλείονται, αλλά θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί στο κείμενο σε σχέση με τη συμπληρωματικότητα, συνέργεια ή συνδυασμό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ε, αποσαφηνήσεις δηλαδή η συνδυασμο θεωρω οτι θα πρεπει να γινουν ορισμενες αποσαφηνίσεις, δηλαδη η παρουσιαση δεν με πίθη, όπως έχει και τέλος από ό,τι άκουσα από τα συνοδευτικά λόγια για το πρόγραμμα, δηλαδή καταπολέμηση της ε, και δημοκρατικές αρχές, δείχνουν από τη φύση τους ότι πραγματικά είναι εντελώς αναγκαίο το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στις ε, διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών. Μπορείς να μεταφέρεις το μήνυμα ότι και εμείς δεν κατανοούμε αυτή την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ DG Home και DG Just και ότι είμαστε πεπισμένες καθόλου ότι είναι ο σωστός δρόμος αυτός ο οποίος επιτρέπει να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε για ένα εύχριστο ολοκληρωμένο πρόγραμμα και ιδίω ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων, διότι υποτίθεται ότι εξυπηρετεί του πολίτε και δεν επιτρέπεται να του προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση με τον περίπλοκο χαρακτήρα του. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο αν θες μπορεί να μεταφέρει. Ευχαριστούμε και όπω είπα καλή επιτυχία στη διαπραγματεύση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, βέβαια έχουμε ήδη σημαντική καθυστέρηση, θα προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε. Ερχόμαστε στο υπαριθμό 10 της ημερησίας διατάξεως, όπου προβλέπεται μελέτη του Policy Department, παρακαλώ ησυχία, γιατί όταν αποχωρείτε προκαλείται πάντα τόσο θόρυβο. Ε, Πρόκειται λοιπόν για την παρουσίαση μελέτη του Policy Department με τίτλο προ ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κινητικότητα στον πολιτισμό». Έχει κέρια σημασία για μας στο νέο μας σχεδιασμό για τον πολιτισμό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου Πολιτισμού, διότι η κινητικότητα των καλλιτεχνών θεωρείται παράγον κλειδί για την βελτίωση της ε, κοινωνικής συνοχής και ως σημαντική συμβολή και για την πολιτιστική διπλωματία. Μήπως σας ενοχλώ εσάς που συζητείτε εκεί κάτω. Η καλλιτεχνική κινητικότητα, η δημιουργική και καλλιτεχνική κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ευτυχώς λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη περισσότερο την προσοχή και της πολιτικής στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη για να προχωρήσει και το νέο πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέπει νέα μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας των καλλιτεχνικών δημιουργών. Χωρίς λοιπόν πολλά λόγια, να δώσω το λόγο στις προσκεκλημένες μας που είναι η κυρία Κλιμεντίνη Ντομπεφ και η κυρία Θεοδόρα Πλετόσου από την ΚΕΑ European Affairs. Είμαι βεβαία ότι θα μας εξηγήσουν οι δύο κυρίες περί τίνος πρόκειται. Σας παρακαλώ ωστόσο να είστε συντομότατες διότι έχουμε ήδη υπερβεί τα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται και γι' αυτό να μην επεκταθείτε σε παραπάνω από 10 λεπτά. Και βεβαίω θα λάβετε το λόγο με την σειρά που εσεί επιθυμείτε. Ορίστε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Είμαι ε, η Κλεμαντίν Ντεμπεφ από την KEA European Affairs. Θα σας μιλήσω για τους στόχους της μελέτης και τη διάρθρωση της έπρεπε να δούμε ποια ε, είναι τα στοιχεία κινητικότητας των ε, επαγγελματιών στην Ευρώπη για να δούμε ποιος είναι ο στόχος και τα χαρακτηριστικά της κινητικότητας καθώς και τα βασικά προσκόμματα προς την ε, κινητικότητα των επαγγελματιών. Επίσης, εκτιμήσαμε το, τη νέα πρόταση ε, δημιουργώντας την Ευρώπη ως προς τη διάσταση κινητικότητας σε ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδότηση για να δούμε ποια είναι μια ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Έχουμε μια ομάδα εργασίας η οποία ξεκίνησε το 2011 και έχουμε ορισμένες συστάσεις σε σχέση με την ε, πλαισίωση της κινητικότητας στα πλαίσια του πιδελταπή. Η μελέτη έδειξε τη σημασία της κινητικότητας για όλους τους τομείς επαγγελματιών, διότι η κινητικότητα τους επιτρέπει να ανταλλάξουν γνώσεις ανά την Ευρώπη και αυτή η κινητικότητα όπως την ορίζουμε είναι η διασυνοριακή μετάβωση από μία χώρα στην άλλη δηλαδή έχει μία καθαρά χρονική διάσταση σε σχέση με την εργασία στις ε, διεθνείς αγορές. Μπορεί κανείς να εμπλουτίσει την επαγγελματική του πείρα και να αναζητήσει και νέες ευκαιρίες. Αυτό το βλέπουμε στα διάφορα σχήματα εργασίας μέσα στα πλαίσια των ε, επιχειρηματικών δυνατοτήτων, άρα η κινητικότητα επιτρέπει την ανάπτυξη της ε, εργασιακής ικανότητας διεθνώς. Είδαμε ότι οι πρακτικές κινητικότητας έχουν άλλες πιο απλές και ευέλικτες μορφές, δεν πρόκειται δηλαδή για μετάβαση ε, έδρας. Υπάρχουν ε, πλήθες προσεγγίσεις και πολύ γνωστικοί τομείς που περιλαμβάνονται και φυσικά υπάρχουν και νέες μορφές κινητικότητας. Αν δούμε το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο βλέπουμε ότι η κινητικότητα δημιουργεί νέες ζωντανές και καινοτόμες κοινωνίες. Γι' αυτό πολλές πρωτοβουλίες κινητικότητας υποστηρίζονται από τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές. Αυτό αφορά το διεθνή διάλογο, διαπολιτισμικές σχέσεις και ανταλλαγές. Είδαμε επίσης ότι η κοινοτικότητα βοηθά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ε, προωθεί την έννοια του ανήκειν και μειώνει τις διαφορές που υπάρχουν ανά την Ευρώπη, όπως θα δούμε λίγο αργότερα στην παρουσίαση. Άρα ε, δεν αφήνουμε κενά στην πολιτισμική διάρθρωση. Είναι ένας καταλήτης για την σύγκληση των πολιτών, κοινά εργαστήρια, εκδηλώσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μία διαφορετική μορφή έκφρασης. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο για να μας μιλήσει για το ρόλο της κινητικότητας σε ευρωπαϊκά επίπεδο. Με βάση λοιπόν αυτές τις διαστάσεις που είπε η συνάδελφος, προσπαθήσαμε να προβούμε σε ένα streamlining στις πολιτικές ε, γειτονίας και εξωτερικών υποθέσεων. Δηλαδή υπάρχει η υπηρεσία διεθνούς ε, ε, διπλωματίας και πολιτισμικής διπλωματίας έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων στα πολιτιστικά. Η COSME είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα και φτάσαμε σε μία σημαντική διάσταση κινητικότητας σε διάφορες διαστάσεις που έχουμε υποστηρίξει οικονομικά. Ορίζοντας 2020 προωθεί την έρευνα και την καινοτομία και έχει προωθήσει προγράμματα και στον τομέα του πολιτισμού. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο συντονισμού μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της κινητικότητας με την, τον, τον ανοιχτό συντονισμό. Μεταξύ 11 και 14 είχαμε τρεις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων που ασχολήθηκαν με ειδικά ζητήματα που άπτονται της κινητικότητας. Τα ευρήματά τους χρησιμοποιούνται και στη δική μας μελέτη για να προωθήσουμε την εργασία σε θέματα κινητικότητας. Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις και τις μελλοντικές δράσεις, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό του Μαΐου του 2018 θέλει να ενισχύσει την κινητικότητα στο, στον πολιτιστικό τομέα και τους ε, τομείς δημιουργίας και υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο για πιλωτικά προγράμματα πολιτισμού στο πρόγραμμα ε, Δημιουργική Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα είναι η πρόταση της Κομισιόν για τη νέα δημιουργική Ευρώπη που θα συζητήσω και αργότερα. Όμως παράλληλα υπάρχουν εμπόδια για την κινητικότητα ως προς κανονισμούς και ένα κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Ο κανονισμός που αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολόγηση δεν έχει τύχει εναρμόνιση στα κράτη-μέλη και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες ε, των καλλιτεχνών και της ε, καλλιτεχνικής κοινότητας. Επειδή υπάρχει μία ενδοδυναμική στη δραστηριότητα του καλλιτέχνη, έχει σημασία το νομικό καθεστώς που τον ε, διέπει και το που απασχολείται. Δεν υπάρχει λοιπόν η κοινωνική προστασία των καλλιτεχνών πάντα. Επίσης υπάρχει φυσικά η, ο αναδιώμενος ε, εθνικισμός στα κράτη-μέλη, το οποίο αποτελεί ένα πρόσκομα στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες επιβαρύνονται φυσικά ε, με μία ειδική φορολόγηση και αυτό αφορά και την κατάσταση μετά το Brexit. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό και ε, τοπικό επίπεδο. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος κατακαιρματισμός. Τα προγράμματα αυτά υπάρχουν περισσότερο στη βορειοδυτική Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν γεωγραφικές ανισότητες που θα πρέπει να αντιπεστούν αντιμετωπιστούν στον ε, πολιτιστικό τομέα. Πολλές φορές εξαρτόμαστε από εθνικές ε, χρηματοδοτήσεις και υπάρχουν και πολιτικά συμφραζόμενα, όπως είπε και η συνάδελφος, μέσα στα πλαίσια του ε, νέου εθνικισμού και γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πληθώρα προγραμμάτων. Υπάρχουν ε, ευκαιρίες ε, για την κινητικότητα, υπάρχει όμως μία ε, διάσπαση αυτών των δραστηριοτήτων, είναι διάχυτες αυτές οι δραστηριότητες, αλλά το κόσμο ή ορίζοντας 2020 δίνει δυνατότητες κινητικότητας οι οποίες όμως δεν είναι ορατές πάντα για τους νέους επιχειρηματίες, γιατί υπηρετούν και την καινοτομία των ΜΜΕ το Erasmus ΣΥΝ δίνει άλλες δυνατότητες κινητικότητας για φοιτητές και νέους επιχειρηματίες κάτω των 30. Σε σχέση με τη διεθνή διάσταση, η εταιρική ανατολική σχέση προβάλλει νέες δυνατότητες, αλλά δεν υπάρχει μία σαφής στρατηγική. Και άρα τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά και δεν υπάρχει συνέχεια των προγραμμάτων σε σχέση ε, με την κινητικότητα στη νέα δημιουργική Ευρώπη. Η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και θα πρέπει να ενισχύσουμε και την διασυνοριακή κυκλοφορία. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα των μελλοντικών πολιτισμικών προγραμμάτων. Δεν ξέρουμε όμως αν θα ταχθεί υπέρ της κινητικότητας όλη αυτή η δραστηριότητα ή εάν θα υπάρχουν ειδικέ δράσεις υποστήριξης όμως. Όπως και να έχει το θέμα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία πλαισίωση της κινητικότητας για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους ε, διαφορετικούς στόχους για ε, τα πολιτιστικά προγράμματα, τους πολιτιστικούς φορείς που θα μπορέσουν να δράσουν ε, διεθνώς. Τώρα η συνάδελφος θα παρουσιάσει το άλλο σκέλος του προγράμματος. Υπάρχουν δύο ε, ομάδες συστάσεων για την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αφιερώνεται στην κινητικότητα στον πολιτιστικό τομέα. Πρώτον, υπάρχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς το οποίο θα είναι συμπληρωματικό σε διάφορα υπάρχοντα ε, προγράμματα που υπάρχουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την στήριξη και την ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα του κλάδου. Αυτό ευθυγραμμίζεται και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και προτείνουμε να κλιμακώσουμε, αν θέλετε, ε, αυτά τα εθνικά και τοπικά συστήματα προκειμένου να ενισχυθεί η, ε, δικτύωση και η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, Θέλουμε καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μέσω ενός διαρθρωμένου διαλόγου που θα γίνεται με τον πολιτιστικό τομέα, προκειμένου να καταργήσουμε ρυθμιστικά εμπόδια. Κάτι που έχουν ήδη κάνει για αρκετά χρόνια ε, επαγγελματικέ ενώσεις στον τομέα του πολιτισμού. Αντίστοιχο έχει γίνει ε, και σε διάφορους, αντίστοιχη έχει γίνει και σε διάφορες προτάσεις κανονισμού. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την κινητικότητα στον πολιτικό τομέα, όχι μόνο γιατί αυτό θα ωφελήσει τον κλάδο που ανέρχεται σε 7,5% του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αλλά και γιατί θα δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία, κάτι που θα μας βοηθήσει και δεδομένων των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ε, για την παρουσίαση της, ε, παρουσία, της μελέτης σας. Σας ευχαριστώ πολύ και ξεκινάμε τώρα με τον, εισηγήτρια, τον εισηγητή μας για το πρόγραμμα Creative Europe. Σίλβια Κώστα, προσπάθησε σε τρία λεπτά, αν μπορείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εκτιμώ τις αξιολογήσεις σας και θεωρώ ότι παρουσιάσατε ένα πανόραμα το οποίο όμως είναι κατακαιρματισμένο. Ε, γι' αυτό δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς φορείς θα πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία πολιτική, δηλαδή το πρόγραμμα της Δημιουργικής Ευρώπης, όπως είδαμε και στην έκθεση εφαρμογής του προγράμματος, και μιλήσαμε και για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κινητικότητας στον πολιτισμό. Ξέρουμε όμως ότι είναι ανεπαρκές, ξέρουμε πώς έχει ο προϋπολογισμός. Πρόκειται λοιπόν για μία εγγραφή που αφορά τον ε, πολιτισμό. Δεν είναι εγκάρσια αυτή η εγγραφή. Έχουμε λοιπόν μία συμπληρωματική εγγραφή στα οριζόντια προγράμματα. Εμείς όμως θεωρούμε ότι για πρώτη φορά γίνεται λόγος ε, για αυτή την εγγραφή στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Όμως το δεύτερο ζήτημα αφορά μια πραγματική πολιτική, ένα πρόγραμμα πλαίσιο που αφορά ευρωπαϊκές και μη χώρες. Εμείς ζητήσαμε από την Επιτροπή προβλέψεις στη νέα στρατηγική για τις διεθνείς διαστάσεις του πολιτισμού και ένα πρόγραμμα κινητικότητας για τις ε, ε, διεθνείς ε, πολιτιστικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να αναλυφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία από εμάς μέσα στα πλαίσια ενός πολιτικού ε, προγράμματος, πολιτιστικού συγγνώμη, προγράμματος ενώ και ενός πιλωτικού προγράμματος. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένα στοιχείο κινητικότητας σε κάθε επιμέρους σχέδιο. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Εσείς θα πρέπει να μου εξηγήσετε πώς το πρόγραμμα θα είναι συμπληρωματικό στα εθνικά προγράμματα. Τέλος, θα ε, θέλαμε να δούμε τι προσκόμματα υπάρχουν. Ε, Σίλβια, έχεις υπερβεί τα τρία λεπτά. Ε, τελειώνω. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει τον καλλιτέχνη και αν υπάρχει διπλή φορολόγηση σε περίπτωση περιοδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ατζέντα πολιτισμού. Ωραία. Θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες. Ποια θα απαντήσει πρώτη. Okay, so about, I will start on the... Uh, Να αρχίσω με την συμπληρωματικότητα με τα τοπικά προγράμματα. Αυτό το σύστημα κινητικότητας θα εφαρμόζεται στο εθνικό επίπεδο από αυτούς τους οργανισμούς. με κάποια εμπλοκή στην διαχείριση ως ε, συμβουλε, παρόχη συμβουλών. με ένα σύστημα επισήμανσης για έμπιστους οργανισμούς υποδοχής. Μπορεί να έχουν ένα είδος ε, σήματος ε, υπεροχής για την κινητικότητα όπως την έχουμε συλλάβει εδώ και για να συμπληρωθεί Mobility Info Points που θα είναι ένα δίκτυο το οποίο παρουσιάζεται σε ορισμένες χώρες μέλη και μάλιστα αυξάνονται οι αριθμοί των χωρών μελών, των χωρών αυτών εν πάση περιπτώσει και βέβαια και σε ορισμένες τρίτες χώρες όπως οι Ενωμένε Πολιτείε. Πρόκειται συχνά για ενώσεις πολύ κοντά στις κυβερνήσεις και διαδίδουν πληροφορίες που απευθύνονται στους επαγγελματίες που θέλουν να μπορούν να έχουν κινητικότητα. Το άλλο είναι η διασύνδεση πόλεων. Πολλές από αυτές είναι δραστηρίες ώστε να λειτουργήσουν ως συγχρηματοδοτούντες εταίροι με την ιδέα όχι να δημιουργηθεί κάτι, να επινοήσουμε εκ νέου τον τροχό, αλλά να βασιστούμε στην υφιστάμενη εμπειρία των πολιτιστικών οργανισμών που μπορούν να στηρίξουν την κινητικότητα. Και τώρα σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πρόγραμμα, λόγω του γεγονότος ότι η κινητικότητα αποτελεί προτεραιότητα μέσα στα πολιτιστικά προγράμματα. Θεωρούμε ότι η κινητικότητα θα συνεχίσει να υποστηρίζεται με διάφορες δράσεις όπως ε, προγράμματα συνεργασίας, στήριξη πλατφορμών και δικτύων αλλά μπορούν να οριστούν και συγκεκριμένες δράσεις θα είναι όμως δύσκολο αυτό από άποψη δημοσιονομική. Γι' αυτό προτείνουμε χωριστές δράσεις για την κινητικότητα ε, πολιτιστικά δημιουργικών επιχειρηματιών και μπορεί να επιληφθεί η ε, αρμόδια γενική διεύθυνση της Επιτροπής. Αυτή είναι η υπόθεση στην βάση της οποίας κινούμαστε. με ειδικό πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ, λέει η Προεδρεύουσα κυρία Τρίπελ. Κύριε κυρία Ζητρογεύσκη, θέλετε το λόγο, ορίστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ομολογώ ότι δεν είμαι ικανοποιημένο διότι Γνωρίζω πώς διαμορφώνεται η ζωή των Ευρωπαίων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών οργανισμών. Μπορώ να χωρίσω το πρόβλημα σε τρεις τομείς. Πρώτον, φορολογία. Τεράστιο πρόβλημα για μας. Ευρωπαίοι καλλιτέχνες εκ διαφόρων χωρών αμείβονται με διαφορετικά ποσά. Παράδειγμα, Πάρτε μια ορχήστρα. Ορχήστρα που αποτελείται από μουσικούς, από προερχόμενους, από ευρωπαϊκές χώρες μέλη. Και ας πούμε ότι έχουν εργαστεί Ιούλιο-Αύγουστο. Κάποιοι θα αμυφθούν, κάποιοι άλλοι θα χάσουν χρήματα. Και αυτό διότι ορισμένοι από τους καλλιτέχνε θα ορίζονται ως καλλιτέχνε, για παράδειγμα Εστονία, Λετωνία. Και τα πρόσωπα αυτά θα μπορέσουν να ε, πέσουν τα έξοδα ταξιδιού και ξενοδοχείων από την αμοιβή του, από, τη φορο, από το φορολογητέο εισόδημα δηλαδή. Άλλοι όχι όμω. Επομένω, αυτοί θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ο ΦΠΑ. Οι κανόνε ΦΠΑ ποικίλουν τόσο πολύ που ίσως είναι δυνατόν να εκπέσουν τον ΦΠΑ, ίσω και όχι. Εξαρτάται πάλι από, από ποιο χώρο προσέσεις Τρίτο, οι καλλιτέχνες ορισμένες φορές λογίζονται ως καλλιτέχνες, άλλες φορές ως επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει νομοθεσία για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει και την καλλιτεχνική δραστηριότητα, ενώ σε άλλες φορές υπάρχει εξειδικευμένη νομοθεσία για καλλιτεχνικές δραστηριότητες, που τους εξαιρεί από την ε, συνήθι φορολογία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι τόσο ποικίλη η κατάσταση ανά την Ευρώπη που αυτό σημαίνει ότι η ελευθερία ε, κυκλοφορίας καλλιτεχνών είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά περιορισμένη. Πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει υπέρ αυτή. βεβαίω και έχουμε το Έρασμό συν για τους κάτω των 30 ετών και είναι ένα θαυμάσιο πρόγραμμα πραγματικά και χάρηκα πάρα πολύ που μπορέσαμε να διπλασιάσουμε τον ε, προπολογισμό του για την επόμενη ε, προγραμματική περίοδο ή οσδήποτε άλλος. Όμως βρίσκεται εκτός του συστήματος των πανεπιστημίων. Εκεί μιλούμε για σημαντικά προβλήματα με τον νόμο, με την φορολογία, με την δήλωση των δραστηριοτήτων των προσώπων αυτών εκτός της χώρας προέλευσής τους. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε σημαντικές αποκλίσεις των ε, ε, φορολογικών καταστάσεών τους ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα να εκπίπτουν ε, δαπάνες μετακίνησης ξενοδοχείων κλπ. Πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Πού θα ασκήσουμε πίεση για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Στην Επιτροπή Πολιτισμού, σε κάποιαν άλλη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή. Ή θα ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα κληθεί μετά να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή. Διότι πρόκειται εν τέλει για την ε, κινητικότητα των καλλιτεχνών. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να επεκταθείτε σε όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια μέσα στο ε, περιορισμένο ε, πλαίσιο αρμοδιοτήτων που σας ανατέθηκε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να επισημάνουμε και εμείς στη μελέτη μας. Συμφωνούμε απόλυτα. Το πεδίο είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένο όσον αφορά τη φερολογία, την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση. Φυσικά ο χρόνος δεν μας επέτρεψε να μπούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να σας παρουσιάσουμε όλες τις, ε, όλα τα στοιχεία, αλλά σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά που αναφέρετε τα εξετάζουμε και εμείς στην ε, δική μας ε, μελέτη επί της ουσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, αρμοδιότητα στον τομέα της φορολογίας. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διευκολύνει, αν θέλετε, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να κινούμαστε προς μια εναρμόνιση των φορολογικών θεμάτων ε, και των θεμάτων που άπτονται της κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από, από αυτή τη συνεργασία και την εναρμόνιση και οι καλλιτέχνε. Υπάρχει μια τέτοια κίνηση σε διάφορους ε, κλάδους ε, εργαζομένων, όχι όμως ιδιαίτερη κίνηση στον τομέα των καλλιτεχνών. Και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσω της μελέτης μας, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα αυτό με τα κράτη-μέλη, με στην ε, Κομισιόν αλλά και εδώ εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Helga Truppel. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπε ο κύριος Σδρογεύσκη είναι ακριβώς αυτό που ε, είναι το αντικείμενο και της μελέτης. Υπάρχει κατακαιρματισμός, υπάρχει έλλειψη πλαισίωσης του ε, καθεστώτος κινητικότητας και έλλειψη συντονισμού. Δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να συντονίσουμε όλα τα εργαλεία και του μηχανισμού που έχουμε στα χέρια μα, να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία ώστε να γνωρίζουν οι πάντε. τι ισχύει. Και μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, είπατε, πόλεις, υπάρχει το κρατικό επίπεδο, υπάρχει το επίπεδο των κρατηδίων στη Γερμανία, υπάρχει το ευρωπαϊκό επίπεδο και χρειαζόμαστε πολύ καλύτερο συντονισμό. Νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι να επινοήσουμε διάφορα καινούργια καθεστώτα και συστήματα, είναι να καθορίσουμε τι ακριβώ θέλουμε να δείξουμε προσήλωση και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τι θα πει η Κομισιόν. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η έλλειψη συντονισμού και κοινή προσέγγιση. Γιατί κάθε μέρα μιλάμε για κοινέ προσεγγίσεις σε διάφορα θέματα, αλλά στον πραγματικό κόσμο, το αναφέρατε κι εσεί, κύριε συνάδελφε, εκτό των πανεπιστημίων, οι καλλιτέχνε πραγματικά δεν ξέρουν τι του γίνεται τι συμβαίνει, τι ισχύει. Και εκεί χρειάζεται να ενισχυθεί η επικοινωνία, ο συντονισμό, η πλαισίωση, να οργανωθούμε καλύτερα για να μπορέσουμε να δρέψουμε και περισσότερου καρπού. Διότι τα πάντα ε, φαίνεται τελικά να τα έχουμε εντάξει στα προγράμματά μα. Δυστυχώ όμω δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να επισπεύσουμε τι διαδικασίε μα, γιατί αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τι ευρωεκλογέ. Γιατί το γνωρίζουμε, όποτε μιλάμε με καλλιτέχνε είναι ότι δεν μας λένε ότι δεν καταλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα συστήματα, οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν, γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει απλούστευση, απλοποίηση, να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα για του ανθρώπου. και αυτό αφορά και την επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Διότι ε, αυτό που θα πρέπει να μα απασχολήσει είναι τι τελικά προσφέρουμε στου καλλιτέχνε στην καθημερινότητά του και στη δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε ε, μπορείτε να πείτε κάτι ακόμη. Το πιλωτικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή pilot project για την κινητικότητα θα δώσει κάποιε κατευθύνσει για το πώ να γίνει καλύτερα η επικοινωνία με του ενδιαφερομένου. Και ένα άλλο που τονίζουμε στη μελέτη μας είναι ότι εξετάζοντας τα πιλωτικά αυτά, θεωρούμε ότι είναι έγκαιρα και ένα καλό πρώτο βήμα. Τους λείπει όμως, τους λείπουν μάλλον οι πόροι για να μπορέσουν να επιτύχουν πραγματικά αποτέλεσματα. Εξετάζουμε και τη χρηματοδότηση που μπορεί να δοθεί σε κάθε μετακινούμενο καλλιτέχνη που είναι πάρα πολύ περιορισμένη και αυτό πρέπει να λυθεί υπόψη λοιπόν δηλαδή ο προπολογισμό που διατίθεται για κάθε, κάθε τέτοιο πρόγραμμα. Και χρειάζεται και εκεί βεβαίω κάποιο συντονισμό. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ, η κυρία Τιμπάτσκα. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις δύο προσκεκλημένες για την ε, παρουσίαση του θέματος. Έχω όμως ερωτήσεις. Έχετε αναλύσει τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην κινητικότητα για τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς και για πρόσωπα από την δημιουργική βιομηχανία, από την βιομηχανία καλλιτεχνικής δημιουργίας δηλαδή. Η δραστηριότητα των Ιταλών και Πολωνών, ας πούμε, έχει μεγάλες διαφορές. Δεν θα μιλήσω καν για ε, Κύπρο ή ε, Μάλτα, όπου η ε, κινητικότητα των καλλιτεχνών εκεί είναι μηδενική σχεδόν. Μπορείτε να σχολιάσετε. Δεύτερο, για το έρασμος συν. Μήπως μπορούμε να αυξήσουμε εκεί το όριο της ηλικία στα 35 από τα 30. Μήπως έτσι μπορεί να επιτευχθεί κάποια συνέργεια μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων και μήπως είναι δυνατόν να ενισχύσει την συμμετοχή των καλλιτεχνών. Σας ευχαριστώ. Λέει Πρόεδρος, ε, ποια από τις δυο σας θα ήθελε να ε, απαντήσει. Θα αρχίσω από το πρώτο ερώτημα. Τα περιορισμένα χρονικά μας πλαίσια δεν ε, διερευνήσαμε τους λόγους ε, των ανισοτήτων ε, μεταξύ κρατών βεβαίως. Αυτό σχετίζεται με τον συνολικό προϋπολογισμό που εγγράφεται για τον πολιτισμό καθώς και την ε, γεωγραφική θέση της χώρας. Αλλά πράγματι η μελέτη μας προσπαθεί να δει τη συνολική εικόνα περισσότερο. Το θέμα που αναφέρεται θα πρέπει να μας απασχολήσει λεπτομερώς. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις ε, για την ε, κινητικότητα και υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης ε, για την κινητικότητα με τη συνέργεια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Γι' αυτό προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια συνολική εικόνα για την Ευρώπη, αλλά σε σχέση με το χρόνο που είχαμε και τους πόρους ε, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τη συνολική εικόνα. Για το Erasmus Sin βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν συνέργειες με τη δημιουργική Ευρώπη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τον αριθμό συμμετεχόντων ή το όριο ηλικίας. Θα πρέπει να δούμε πώς το πρόγραμμα θα ενταχθεί στο επόμενο πι, έτσι ώστε να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Υπάρχουν όμως συνέργειες ως προς το συμπληρωματικό χαρακτήρα αυτών των δύο προγραμμάτων της Δημιουργικής Ευρώπης και του Erasmus Συν. Το Erasmus Συν δίνει αυτή τη δυνατότητα κινητικότητας σε ε, ηλικίε που αφορούν και επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να μπορέσουν να εμβαθύνουν τις δεξιότητες που διαθέτουν και αυτό μέσα στα πλαίσια και της συνέργειας του Erasmus Συν στο επόμενο ΠΔΠ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο πρώτο ερώτημα. Θα πρέπει να δούμε και τη δραστηριότητα των εθνικών οργανισμών. Ας πούμε το ΓΚΕΤΕ ή το Γαλλικό Ινστιτούτο, το αντίστοιχο της Ιταλίας ή ε, της Ισπανίας το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μεγάλες οργανώσεις, μεγάλοι οργανισμοί μάλλον, που ε, προωθούν την ε, κινητικότητα. Αυτά τα Ινστιτούτα όμως έχουν ε, διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με τη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Η Julie Ward έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η μελέτη αυτή και αναδεικνύει πράγματα που τα γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Εγώ εργαζόμουν στον πολιτικό τομέα και είναι αλήθεια όλα αυτά που λέτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει πραγματικά να κάνει κανεί τεράστια προσπάθεια όταν, αν είναι, όταν ως καλλιτέχνης αν θέλει να παρουσιάσει το έργο του διασυνοριακά με άλλους ε, συνεργάτες ε, στην Ευρώπη δουλεύουν εξαιρετικοί άνθρωποι. Είναι εδώ και μαζί μας η κυρία Χριστοφόρου από ε, μια Βρετανική οργάνωση η οποία πραγματικά έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια ε, για τον συντονισμό και τη συνεργασία καλλιτεχνών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και από τις γειτονικές μας χώρες. Νομίζω, ξέρετε, οι, οι καλές τέχνες και ο πολιτικός τομέας ε, επιδεικνύουν μια, μια αξιέπαινη ε, ανθεκτικότητα ε, και την επέδειξαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί, πρέπει να το γνωρίζει η Κομισιόν. Δεν είναι κάποια, κάποιος περιφερειακός κλάδος που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική επιτυχία μας. Είναι ε, θεμελιώδους, κεφαλαιόδους σημασίας ο ρόλος του πολιτισμού, για την ευζοία της Ευρώπης, για την, για την ζωή των τοπικών κοινωνιών, για τις κοινωνίες εν γέννη. Νομίζω ότι λοιπόν μπορεί αυτός ο κλάδος απλά να περιορίζεται και η συζήτηση γύρω από αυτόν εδώ στον δικό, στη δική μας επιτροπή που είναι, είμαστε και καθήλυνα αρμόδια. Πρέπει να αναγνωρίζουμε αυτά τα θέματα και στις άλλες επιτροπές, διότι αν, υπάρχει προβλήμα, αν υπάρχουν προβλήματα στον πολιτικό κλάδο, ε, αυτό δημιουργεί κόστος και για την οικονομία μας και για την κοινωνική συνοχή μας, διότι οι καλλιτέχνες πολλές φορές κάνουν αυτήν τη δουλειά, φέρνουν μαζί τον κόσμο στον ίδιο χώρο, ε, δουλεύουν με πρόσφυγες, δουλεύουν με ανθρώπους αποκλεισμένους, περιθωριοποιημένους στις κοινωνίες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα να αποσταλεί και σε άλλους. Και να μην μένουμε εδώ στου τέσσερις τείχου επιτροπή Επιτροπής μας και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή που ακούστηκε για τη διεύρυνση του προγράμματος Erasmus+. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ιδίως για τα φεστιβάλ ε, τα φεστιβάλ αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αν θέλετε διότι συνιστούν μια δημόσια παρουσίαση του, της κινητικότητας αλλά θα έχουν ε, πολλά προβλήματα τα φεστιβάλ το επόμενο διάστημα ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά το Brexit ε, τα φεστιβάλ και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου θα αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα εξαιτία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σύντομα, ναι. Θα είμαι σύντομη. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση Φεστιβάλ ε, κινητοποιείται πολύ για το θέμα αυτό, τη κινητικότητα δηλαδή, όπως είπατε και εσείς και το τονίζουμε και εμείς στη μελέτη μας, ιδίω η βρετανική αποχώρηση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στον ε, καλλιτεχνικό κλάδο και βέβαια και ιδιαίτερα για τα φεστιβάλ και τη δυνατότητα υποδοχής ε, αλλοδαπών καλλιτεχνών η εταίρα των προσκεκριμένων. Να προσθέσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι ο τομέας των καλλιτεχνών, της καλλιτεχνικής δημιουργίας δηλαδή, είναι οριζόντιος και υπησέρχεται σε πολλούς άλλους. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι οι ευκαιρίες που δίνονται είναι αρκετά κρυμμένες σε άλλες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τα γνωρίζουν αυτά οι καλλιτέχνες ας πούμε, στο κόσμο ή στο, Ευρω... ορίζον 2020. Και λίγες δημόσιες διαβουλεύσεις γίνονται για το μέλλον των δραστηριοτήτων αυτών και δεν θίγουν τον καλλιτεχνικό δημιουργικό τομέα και αυτό είναι κρίμα γιατί ε, εκεί αυτός μπορεί να βοηθήσει στην ε, κινητικότητα των καλλιτεχνών και θα είναι σωστό να περιληφθούν να περιληφθεί ο τομέας, ο κλάδος σε μελλοντικέ δημόσιες διαβουλεύσεις. η πρόεδρος κυρία Κάμερ Έβερτ, Σας ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά οφείλω να ομολογήσω ότι σε ό,τι αφορά την ε, επέκταση του ορίου ηλικία για το έρασμο δεν είμαι πολύ βεβαία διότι αφενός ζητούμε περισσότερα κονδύλια πρέπει ωστόσο να προσέξουμε να μην το ε, παραεπεκτείνουμε το πρόγραμμα ώστε τελικώς δεν φτάνουμε στους παραλήπτες και δικιούχους που επιθυμούμε να φτάσουμε και να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες για ανταλλαγές καλλιτεχνών. Σας παρακαλώ τώρα πολύ σύντομα διότι έχουμε πάλι ξεπεράσει το χρόνο μας και θα ήθελα να ακούσω και την κυρία Γκέσλερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Μπίλτ, ορίστε παρακαλώ. Εντάχει καλημέρα σας ε, κυρίες μου. Η δική σας υποστήριξη έχει ως εξή σελίδα 33 λέτε ότι η αύξηση του εθνικισμού, ο ευρωσκεπτικισμός και η ξενοφοβία έχουν επίπτωση στην κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων. Καταρχήν, αν ε, υπάρχει κάτι που τροφοδοτεί την, ε, τους εθνικισμούς είναι ότι έχουμε ξεχάσει τον κόσμο, έχουμε ξεχάσει τους πολίτες ως προς τον εθνικισμό θα υπάρχει όσο υπάρχουν και τα έθνη. Η έκθεσή σας ε, θέλει την εξάλληψή του γιατί λυπόσαστε για το γεγονός ότι υπάρχουν σύνορα που πρέπει να διαβεί ε, κανείς. Εάν θέλετε να κάνετε πολιτική, τότε να σας εκλέξουν καλύτερα. Θα ήταν πιο απλό. Φαίνεται ότι αυτό που λέτε, αυτά που λέτε έχουν επιπτώσεις. Μα αυτά είναι οι προσωπικές σας απόψεις δεν νομίζω ότι τη σημερίζονται πολύ. Μιλήσατε για την Ουγγρική Ακαδημία Τεχνών. Είπατε ότι είναι ένας οργανισμός πιστός στο έθνος και λέτε ότι η Ουγγρική κυβέρνηση κατασπαταλά τα χρήματα αυτού του οργανισμού. Δηλαδή, τι λέτε, ότι οι Ούγγροι δεν θα έπρεπε να ε, προασπίζονται ή να υπερασπίζονται τον πολιτισμό τους. Μη συντάσετε εκθέσεις. Πηγαίνετε να βρείτε τον κύριο Σόρος, ο οποίος θα ήθελε να χρηματοδοτήσει έναν πολιτισμό όπως αυτόν που εύχεστε εσείς. Um, Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι η έκθεσή μας αντιθέτως υπερασπίζεται την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης και θέλει να προστατεύσει αυτήν την πολυμορφία που ε, υπάρχει στους διάφορους πολιτισμούς. Αυτό που ζητούμε είναι να υπάρχει μια ανταλλαγή μεταξύ των διαφόρων ταυτοτήτων και πολιτιστικών υποβάθρων ακριβώς για να μπορούμε να αναδείξουμε τις πολιτιστικές διαφορές και ιδιαιτερότητες και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ. Ε, Απλώ να σα υπενθυμίσω ότι και οι καλλιτέχνε είναι Ευρωπαίοι πολίτε, λέει η πρόεδρο. Μπάρμπαρα Γκέσλερ. Όσο πιο σύντομα μπορεί σε παρακαλώ, ξέρω είναι δύσκολο. Ευχαριστώ που μου δίνεις το λόγο. Σας ευχαριστώ καταρχάς ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ανέθεσε την εκπόνηση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη η παρουσίαση αυτής της μελέτης σε σχέση και με τα όσα κάνουμε κατά τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Πράγματι λοιπόν θεωρούμε ότι η κινητικότητα είναι μια διάσταση που υπάρχει ε, έχει ενταχθεί σε όλες τις διαστάσεις του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Υπάρχει ήδη αυτή η κινητικότητα, ήδη. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες μας και την ε, διασυνοριακή, αν θέλετε, απήχηση των καλλιτεχνών. Αυτή άλλωστε είναι και η προστιθέμενη αξία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγκυται στην κοινοτικότητα. Αυτό αναδεικνύει και η μελέτη. Αλλά ε, όπως λέει και η μελέτη ε, υπάρχει ανάγκη ε, να με συγκεκριμένο τρόπο να επεξεργαστούμε και να ενισχύσουμε την κινητικότητα και των καλλιτεχνών με εξειδικευμένο τρόπο. Και αυτό η ανάγκη αυτή ανεδείχθη νομίζω εξαιρετικά από τη μελέτη. Συμφωνούμε πράγματι υπόρρητα στην ε, δημιουργική Ευρώπη ε, η κινητικότητα υπάρχει ως οριζόντια διάσταση. Τις επόμενες ε, δύο εβδομάδες θα καταλήξουμε και στον διαγωνισμό, στα αποτελέσματα του διαγωνισμού που διοργανώσαμε. Λάβαμε πολύ καλές προτάσεις. Το πρώτο βήμα σε αυτό το πολιτικό πρόγραμμα που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ε, και χάρη στη συμβολή του Κοινοβουλίου είναι και η εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα και πραγματικά, όπως υπόθηκε σήμερα στη συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί η ιδέουσα σημασία σε αυτή την πλατφόρμα. Πρέπει να ενισχυθεί η επικοινωνία. Όλοι το τονίσατε αυτό στις τοποθετήσεις σας. Και τρίτον, θα περάσουμε σε μια πειραματική φάση στην οποία θέλουμε να δοκιμάσουμε και να ελέγξουμε τι μορφή θα μπορούσε να έχει αυτή η πλατφόρμα, αυτή η επικοινωνία. Ε, θα πρέπει, επειδή δεν υπάρχει μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο, πρέπει να δούμε πώ ακριβώ θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο μηχανισμό, ποιε θα είναι, ποιες θα είναι οι ομάδε στόχοι, ώστε στο τέλο τη επόμενη χρονιά να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε συστάσει για τη μετουσίωση όλων αυτών που θα έχουμε διαπιστώσει σε απτά μέτρα στο πλαίσιο του Δημιουργική Ευρώπη. Κάτι για το χρονοδιάγραμμα να σας πω. Βρισκόμαστε βεβαίως σε διαδικασίες συζητήσεων με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να καταργήσουμε τα εμπόδια στην κινητικότητα με τα κράτη-μέλη και όλα αυτά βεβαίως θα συνοδευτούν και από χρηματοδοτική στήριξη από πλευράς Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε και άλλες αφορμές πολλές για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο προσκεκλημένες για την παρουσία σας εδώ σήμερα, για την παρουσίαση της μελέτης που νομίζω μας δίνει σημαντικές διαστάσεις για την παραπέρα εργασία μας και για το πρόγραμμα καλλιτεχνική, ε, Δημιουργική Ευρώπη, αλλά και για τον περαιτέρω προγραμματισμό των δράσεων στον τομέα του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. So, για να προχωρήσουμε τώρα, μάλλον πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, με μεγάλη χαρά απευθύνω το καλό ορίσατε σε 16 φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου της Φεράρα. Έχετε έλθει εδώ μετά από πρόσκληση της ε, φίλης μας Σίλβια Κώστα. Ελπίζω να συλλέξετε ενδιαφέρουσες εμπειρίες από την παραμονή σας εδώ. Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως του σημερινού πρωινού και είναι μεγάλη η χαρά που με διακατέχει που μπορώ να σας παρουσιάσω τους νικητές των τριών πρώτων βραβείων του βραβείου Καρλομάγνου. Τους τρεις πρώτους νικητές δηλαδή του βραβείου Καρλομάγνου. Ε, είναι μια θαυμάσια ε, συνήθεια πλέον, ε, παράδοση που έχουμε τους τρεις πρώτους νικητές από την ε, εκδήλωση αυτή και δίνουμε την ευκαιρία στα πρόσωπα αυτά να παρουσιάσουν τα projects τα οποία έχουν εργαστεί και για τα οποία βραβεύτηκαν και τουλάχιστον η εμπειρία των τελευταίων ετών είναι ότι ο ενθουσιασμός τους για την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές ιδέες είναι και μεταδοτικό. Έχουμε λοιπόν τους εκπροσώπους των τριών ομάδων, των τριών τριών ομάδων από Πολωνία, Ιταλία και Μάλτα. Πολωνία, Ιταλία και Μάλτα. Αφενός ο Τόμας Τόμαλικ που θα παρουσιάσει το project Walkation από την Πολωνία. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος ο Τόμας ε, περί τίνος πρόκειται. Το δεύτερο βραβείο κατέκτησε η Τζουβενίλια από την Ιταλία και θα το παρουσιάσει ο Μίρκο Γκρανιάτο. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Never Arrive 2 από τη Μάρτα που παρουσιάζει η Φαρά Αμπτουλαχή Αμπτή. Και τα τρία αυτά πρόσωπα θα μπορέσουν να παρουσιάσουν το project το οποίο βραβεύτηκαν ε, δεν ξέρω ποιο ή ποια θα αρχίσει. Έχετε 7 λεπτά ο καθένας και μετά θα έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Ποιο θα ήθελε να αρχίσει. Θα θέλατε εσεί, Πολύ ωραία. Αρχίζετε λοιπόν εσείς με το, ε, ε, πρόγραμμα, με το ε, πρόγραμμα, το έργο Never arrive 2 από τη Μάλτα. Έχετε 7 λεπτά. Είμαι η Φάρα, ε, κατάγομαι από τη Σομαλία και ζω στο Βερολίνο. Αυτά είναι τα γερμανικά μου. Μόλις ε, έχω μετακομίσει στη Γερμανία και μαθαίνω γερμανικά. Λοιπόν, το project μου έχει τον τίτλο Never Arrive To. Αποτελεί μια συνέχεια της αυτοβιογραφίας μου την οποία ξεκίνησα να γράφω το 2013 και εκδόθηκε το 2016 ως ε, διεμφυλική πρόσφυγας που εγκατέλειψα τη χώρα μου για λόγους ασφάλειας προσωπικής προφανώς για να έρθω στην Ευρώπη, για να μπορέσω να ζήσω τη ζωή μου και κάνοντας αυτό το δύσκολο ταξίδι από την υποσαχάρια Αφρική, περνώντας την έρημο, τη Μεσόγειο θάλασσα, φτάνοντας στη Μάλτα με βάρκα το 2012 περνώντας από τη διαδικασία κράτησης, ε, αίτησης ασύλου, έζησα τέσσερα χρόνια εκεί. Προσπάθησα να ενταχθώ στην κοινωνία, να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Ξέρετε ότι η μετανάστευση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη, για ολόκληρο τον κόσμο. Και έτσι θέλησα να, να γράψω ένα βιβλίο που θα ε, διηγείται με θετικό τρόπο το ταξίδι της μετανάστευσης. Να ε, αντικρούσουμε αυτήν την εικόνα του πρόσφυγα που έρχεται να καταστρέψει τον πολιτισμό της Ευρώπης. Ήθελα να μιλήσω για τα οράματά μου, για τις φιλοδοξίες μου, για τα ε, όνειρά μου, για τους ανθρώπους που απλώς θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους ε, κατάφερα λοιπόν ε, στη διαδικασία αυτή ε, με το βιβλίο να ταξιδέψω σε διάφορες χώρες. Προλόγησε και το βιβλίο μου η πρώην Επίτροπος Ιστορικών Υποθέσεων και σκοπός μου είναι να ενθαρρύνω τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, να τους πω ότι το ταξίδι θα είναι δύσκολο, αλλά θα, θα στεφτεί με επιτυχία στο τέλος. Το Never Arrive 2 ε, είναι λοιπόν μια, ένα εγχείρημα, μια προσπάθεια να ενθαρρύνουμε τόσο τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, αλλά και τους ανθρώπους που ζουν στις χώρες υποδοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί μια ανοιχτή συζήτηση για τη μετανάστευση, για τις τοπικές κοινωνίες, για τις κοινότητες, για να αρθεί ο φόβος που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι άπαξ και δημιουργηθεί αυτός ο σύνδεσμος, αυτή η επικοινωνία, είναι πιο εύκολο να καταργηθούν εμπόδια, μπορούν άνθρωποι να ε, ε, ζήσουν μαζί, να συζητήσουν ε, να ξεπεράσουν όταν δηλαδή οι άνθρωποι που τους έχουν βομβαρδίσει με εικόνες ανθρώπων που καταφτάνουν σε πλοιάρια στις ακτές τους όταν, τους, ε, όταν γνωρίζει κανείς, ε, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει πραγματικό πρόσφυγα και μετανάστη, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ σα είπα ότι αν δοθούν ευκαιρίε στους μετανάστε, εγώ ζω εδώ και έζησα τέσσερα χρόνια ε, στη Μάλτα, τώρα είμαι στο Βερολίνο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί από εμά που καταφέρουμε, γινόμαστε νοσοκόμε, γιατροί, αν μα δοθούν οι ευκαιρίες. βεβαίω από την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που λόγω των δυσκολιών και των κακουχιών καταλήγουν στην εγκληματικότητα, στο περιθώριο της κοινωνίας. Και εκεί επικεντρώνεται η ακροδεξιά. Αυτά τα, αυτές τις εικόνες προσπαθούν να, ε, να προβάλλουν στους ψηφοφόρους τους. Δεν, ε, δεν προβάλλουν μετανάστες πρόσφυγες που μπορεί να είναι make-up artists ας πούμε ή που μπορεί να ασχολούνται με τη μόδα ή με άλλους καλλιτεχνικούς τομείς. Αυτό που θέλω λοιπόν να ενισχύσω είναι αυτή η εικόνα ότι ότι η ζωή μας αφορά την ταυτότητα, την αγάπη, την, την δυνατότητα να ζήσεις την δική σου αλήθεια αν θέλει. να μπορεί να πει ένας άνθρωπος ότι αυτό που αντιμετωπίζω στη ζωή μου δεν είναι για εμένα. Γι' αυτό και επέλεξα αυτόν τον ε, τίτλο, το Never Arrive. Ε, αυτό ήταν και αυτό που μου έλεγε η μαμά μου. Να μην αφήνω τους άλλους ανθρώπους να προκαθορίσουν το δικό μου, τον δικό μου προορισμό. Αφού λοιπόν βρέθηκα στην Μάλτα και διαπίστωσα ότι δεν χωρούσα σε αυτόν τον τόπο, αποφάσισα να φύγω. Είδα τη Μάλτα, ήταν αρκετά περιορισμένα τα πράγματα που μπορούσα να κάνω εκεί, γι' αυτό και αποφάσισα να πάω στο Βερολίνο και εκεί μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Να μην αφήνετε να σας κλέψουν τα, τα όνειρά σας, τις φιλοδοξίες σας. Μπορείς να πάρεις τα κοσμήματά μου, τα υπάρχοντά μου, γιατί αυτό μου συνέβη εμένα. Άφησα πίσω μου όλα μου τα υπάρχοντα. Όμως επιδίωξα να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και νομίζω ότι αυτό, αν κάνεις αυτό, αυτό θα σου δώσει τη δυνατότητα να ξαναγοράσεις όλα αυτά τα υλικά αγαθά που αναγκάστηκες να εγκαταλείψεις και να αφήσει πίσω σου. Κοσμήματα, σπίτια, ό,τι θέλεις. Αυτό λοιπόν θέλω να είναι το μήνυμα αυτή της παρουσίας μου εδώ και του βιβλίου μου. Ε, θα ήθελα φυσικά και το δεύτερο βιβλίο μου να μεταφραστεί και στα γερμανικά, που είναι πλέον η δεύτερη πατρίδα μου. Μου λένε οι άνθρωποι ότι λες στους ανθρώπους να μην, να μην φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει κάθε άνθρωπος και οι μετανάστες να έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αυτό μου έδωσε και εμένα το Βερολίνο στην παρούσα φάση της ζωής μου. Αυτό μου έχει δώσει το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Never Arrive. Και αυτό επιδιώκω και ελπίζω και για όλους τους άλλους ε, συνανθρώπους μου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πραγματικά εντυπωσιακή παρουσίαση του project σας και θα συζητήσουμε ε, μόλις ακούσουμε και τις τρεις παρουσιάσεις, τις άλλες δύο ακόμη δηλαδή. Ερχόμαστε στο δεύτερο βραβείο, Τζουβενίλια, από την Ιταλία, που την παρουσίαση θα κάνει ο Μίρκο Γκρανιάτο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι κάτι το μαγικό. Πριν μιλήσω για το Γιουβενίλια και σας δείξω ένα βίντεο, θα ήθελα να αρχίσω με τον Ουμπέρτο Βελιμπέρτη που έγραψε ένα βιβλίο για τους νέους. Ο Βελιμπέρτη λέει ότι Εάν ο άνθρωπος ε, θέλει να φτάσει στη λογική, ε, λαμβάνοντας υπόψη τον ηχηλισμό της εποχής, ε, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει μία πολιτισμική ανησυχία, όπως είχε πει και ο Γκέτε. Και φυσικά το να υποφέρουν οι νέοι σημαίνει δυστυχώς ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχει σύγκληση για τους ε, νέους. Ε, ο Γκαλιμπέρτη έγραψε ε, την ίδια εποχή που εμφανίστηκε και το βραβείο του Καρλομάγνου. Πρόκειται για ένα βίντεο που διαρκεί ένα λεπτό. Μετά τη θέσπιση του βραβείου του Καρλομάγνου. No. Ok. το βίντεο προέβλεπε και μουσική. Ε, η μουσική ήταν ε, του Γκρίγκ. Ε, δυστυχώς ξέρω ότι υπάρχει και στενότητα χρόνου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Φαίνεται ότι το Γιουβενίλια διαθέτει πολλά χρήματα, έχει κονδύλια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, θα ήθελα να σπάσουμε στερεότυπα. Εμένα μου αρέσει πολύ κλασική μουσική. Ο πατέρας μου ήταν πυροσβέστης, είναι πυροσβέστης και η μητέρα μου ασχολήθηκε με τα οικιακά. Η μουσική είναι για όλους, δεν είναι για ε, μερικούς. Όταν ε, ο Μάριο τραγουδάει «Ελουτσέβαν Λεστέλε», όταν ε, τραγουδάει Κάρμεν, όλοι ε, βρισκόμαστε σε μία κατάσταση ε, ευθυμίας. Εμείς θέλουμε ως εθελοντές να φέρουμε σε επαφή νέους από ολόκληρη την Ευρώπη για να ζήσουν την εμπειρία του θέατρου όταν ήμουν 16 ετών πήγε ένα θέατρο μόνος μου, δεν με ε, ακολουθούσε κανείς. Η κλασική μουσική όμως έχει μία μεγάλη εσωτερική δύναμη και θεωρώ ότι θα πρέπει να συμμεριζόμαστε, σε αυτές τις, ε, ε, να συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δυστυχώς δεν με βοηθάει η τεχνολογία Μίλαμε λοιπόν για νέους Ευρωπαίους και φίλους της όπερας. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τις πόρτες του θεάτρου σε όλους. Μπορεί κανείς να συμμετέχει σε μία οργάνωση, μπορεί να είναι νεοφώτιστος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να πρόκειται για μία εμπειρία που μοιραζόμαστε όλους. Ε, ένας νέος Άγγλος μου έλεγε ότι η όπερα είναι σαν να πηγαίνει κανένας σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Το ίδιο συμβαίνει και με την όπερα. Είναι όπως ένας αγώνας ποδοσφαίρου που μιλάει σε πολλούς. Στο τέλος όλοι χειροκροτούμε. Εμείς τα, στη Γιουνβενίλια θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες. Το θέατρο δυστυχώς ε, έχει μεγαλύτερη ε, κοινωνική στρωματοποίηση, αλλά στη Γιουβενίλια δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Μπορούμε να πάμε στις πλατείες, στα θεωρία, οπουδήποτε μέσα στα πλαίσια ε, ενός πολύ περιορισμένου προϋπολογισμού. Εμείς ε, μιλάμε με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, με τους υπεύθυνους και προσπαθούμε να ανοίξουμε το θέατρο σε όλους, σε μια λογική τιμή, έτσι ώστε οι νέοι να έρθουν στη σκάλα του Μιλάνου και να συμμετέχουν να μπορέσουν δηλαδή να καθίσουν σε θέσεις της πλατείας με 20 ευρώ. Έτσι να μπορέσει κανείς να ανακαλύψει και πόλεις. Το θέατρο είναι ένα άνοιγμα προς τον κόσμο, ο οποίος φαίνεται πολλές φορές απροσπέλαστος. Η Γιουβενίλια προσπαθεί να πλαισιώσει πολλούς νέους ανθρώπους, γιατί πρόκειται για ένα κοινό πάθος για την μουσική. Όταν αρχίζει, αρχίζει κανείς ε, να μιλά για τη μουσική, βλέπουμε ότι υπάρχει μία συμφιλίωση των ανθρώπων. Φτάνουμε σε ένα ε, σχήμα νέων που μπορεί να μεταβεί από το Βερολίνο στη Βαρκελόνη και μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίες. Στο συντονισμό συμμετέχουμε Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, πολλές εθνότητες και υπάρχει αυτή η, τάση που ενώνει τους ανθρώπους. Μπορώ να τραγουδήσω μία άρια του Μότσαρτ στα γερμανικά. Το έχω μάθει. Βλέπετε ότι φτάνουμε από το Όσλο μέχρι το Τεάτρο Μάσιμο του Παλέρμο. Στο Τεάτρο Μάσιμο υπάρχει μία επιγραφή που λέει ότι η τέχνη ανανεώνει τους ανθρώπους και τη ε, ζωή. Εμείς δεν πάμε στην όπερα γιατί θέλουμε να γεμίσουμε ένα βράδυ μας. Συμμεριζόμαστε κοινέ αξίες. Μακρηγορώ, το ξέρω. Το θέατρο είναι ένας μαγικός τόπος γιατί εκεί εργάζονται όλοι από τον τραγουδιστή μέχρι τον υπεύθυνο της ορχήστρας, τον ηλεκτρολόγο, τον υπεύθυνο φωτισμού, τον ε, ξυλογλύπτη, τον μαραγκό, τον σκηνογράφο και όλες τις ειδικότητε. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε αυτόν τον κοινό σκοπό. Πώς συνεργάζονται όλοι για ένα μεγάλο θέαμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτού του θαυμάσιου ε, project και ας έρθουμε τώρα στο πρώτο βραβείο ε, του φετινού ε, κύκλου από την Πολωνία. Walkation. επιγράφεται και θα το παρουσιάσει ο Τόμας Τόμαλικ. Ευχαριστώ, λέγομαι Τόμαλικ και είμαι Πολωνός. και είμαι <clears throat> ακόμα στο Λύκειο, στο Βρότσλαβ. Και είναι μεγάλη χαρά μου που μου επιτρέπετε να παρουσιάσω το project εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω έρχομαι εδώ για πρώτη φορά. Στις αρχές του 2018 υπέβαλα το σχέδιο του Workation για το βραβείο νεολαία του Καρλομάγνου. Κερδίσαμε σε εθνικό επίπεδο. Και να είμαστε τώρα ως νικητές και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας πω τι είναι το Workation. Κάθε χρόνο προσκαλούμε νέους από Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρωμανία και Ιταλία, Ρουμανία και Ιταλία, στο Γκέρδης και στο Σγκόρζελικ. Τα πρόσωπα αυτά έχουν την ε, δυνατότητα να συνεργαστούν, να περάσουν καλά και να μιλήσουν βεβαίω, να συνεννοηθούν μεταξύ τους σε διαφορετικές γλώσσες. Σκληρή δουλειά όμως, αλλά έχει και πλάκα. Και ιδίω όταν ε, αρχίσουν να γνωρίζονται μεταξύ τους. Αυτά γίνονται και σε τοποθεσία ενός πρώην γερμανικού στρατοπέδου συγκέντρωσης από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είχαμε δύο ομάδες, αρχαιολόγους και καλλιτέχνες. Οι αρχαιολόγοι προχώρησαν σε ανασκαφή, όπου βρήκαν ψηφίδες ντόμινο και κέρματα η άλλη ομάδα έφτιαξε μάσκες από μέταλλο με, υπό την καθοδήγηση ε, επαγγελματία το, αυτό το 2017. Το 2016 η ομάδα των αρχαιολόγων ανεκάλυψαν διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Οι δε καλλιτέχνες έφτιαξαν εγκαταστάσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας από κλαδιά κλπ. Μιλήσαμε για, την, για τις μνήμες. Ε, αναρωτηθήκαμε αν υπάρχει κάτι που να είναι ευρωπαϊκή μνήμη. Τέτοιες συναντήσεις με τέτοιες εθνικότητες καταλήγουν στο ότι χρειάζεται να μπορούμε να διδαχτούμε από την ιστορία και να μπορούμε να σχεδιάσουμε το κοινό μας μέλλον. Βλέπετε εδώ και φωτογραφίες από τις δραστηριότητες αυτές. Στο τέλος του project, του work camp, έγινε και απαγγελία ποιησης. Και είδαμε και προσκαλέσαμε και ντόπιου από τον Γκέρλις και τον Σκόρζελεκ σε μια τελετή και αυτά κλείνουν και με, και μια συναυλία. Το έργο μας, ...Walkation δηλαδή, σημαίνει και συνεργασία αλλά και κοινή διασκέδαση, ε, οργάνωση κοινού χρόνου, ε, με παιχνίδια, με το να ε, εξερευνήσουμε το περιβάλλον του χώρου αυτού του στρατοπέδου συγκεντρώσεως. Βλέπουμε και τα όσα συμβαίνουν εκεί γύρω και στην ουσία αναβιώνουμε την ιστορία. Ο χρόνος που μου διαθέσατε ήταν λίγος, προσπάθησα ωστόσο στο περιορισμένο αυτό χρόνο να σας εξηγήσω τι είναι το workation. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα. Σας είπα όμως αυτά που εγώ θεωρώ πιο σημαντικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτού του εντυπωσιακού και πολύ σημαντικού project. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν μπορεί να διαμορφώσει και το μέλλον του. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε και στην σημερινή γενιά, στη νέα γενιά, ε, πόσο ε, άσχημη ήταν η κατάσταση στην Ευρώπη πριν από, στο όχι και πολύ απότερο παρελθόν και ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει ποτέ ξανά να συμβούν στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι τα τρία αυτά project με διαφορετικό τρόπο το καθένα απέδειξαν πόσο δημιουργικοί μπορούν να είναι οι νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη με πόση θέρμη εργάζονται και οι νέοι άνθρωποι για να βελτιώσουν λίγο-λίγο την Ευρώπη, πώς μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν στην ε, αλληλοκατανόηση μεταξύ των διαφόρων ε, πολιτισμών, των διαφόρων τρόπων ζωής που υπάρχουν πώς μπορούν να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων για όλα αυτά τα θέματα, πώς μπορούν να αναδείξουν τις διαφορές για να γεφυρώσουν τους λαού και όχι για να ανεγείρουν τύχη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνετε. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας να περάσουμε στη συζήτηση, να δώσω το λόγο στην ε, Σαμπίνε Φερχάιν από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Καταρχά θέλω να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα εδώ και για την παρουσίαση του έργου σα. Είχα την τιμή άλλωστε και στην, ε, να είμαι και στην ε, απονομή του βραβείου Καρλομάγνου στο Άχεν, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Και πρέπει να πω ότι όλοι οι νικητές του βραβείου με εντυπωσίασαν βαθύτατα. Ε, πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της ε, Κριτικής Επιτροπής που κλήθηκε να ε, διαλέξει τρία ε, project για την βράβευση ακριβώς γιατί υπήρχε μια τεράστια ποικιλομορφία που την είδαμε και σήμερα εδώ στους βραβευθέντες. Υπάρχει μια πλειάδα τρόπων με τον οποίο μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ζήσει την Ευρώπη, την ενωμένη Ευρώπη και πώς μπορεί να συμμετάσχει και να συνεισφέρει και εκείνος στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ιδιαίτερα με εντυπωσία, δεν θέλω ε, να είμαι άδικη, αλλά πραγματικά με εντυπωσίασε πολύ αυτό το project γύρω από την όπερα. Πώς μπορούμε δηλαδή να καταστήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά προσβάσιμη στους νέους ανθρώπους και σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η κλασική μουσική ε, κάποτε ε, ε, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν φέουδα και βασίλεια συνέδεαν, συνέδεε η μουσική, η κλασική μουσική τους διάφορους λαούς, τις εθνότητες της Ευρώπης και γι' αυτό είναι και εξαιρετικό εργαλείο <laughs> το να Υπάρχει η, δυνατότητα αυτή να αναδεικνύουμε την μουσική ως εργαλείο που μπορεί να σταθεί απέναντι στον εθνικισμό. Αυτό είναι και πολύ σημαντικό και ως προς αυτό που κάνει το workation, πώς μπορούν δηλαδή οι νέοι άνθρωποι να μάθουν τι τελικά ήταν εκείνο που χώρισε τους λαούς της Ευρώπης στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τι τελικά όμως κατάφερε και τους ένωσε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό να, να, και οι δύο διαστάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα της, ε, την Ευρώπη. Και σε αυτό πραγματικά ρόλο, σε αυτό ρόλο έχουν να παίξουν και οι μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να δείξουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε σε εκείνους τι τελικά είναι η Ευρώπη, ποιες είναι οι αξίες της και νομίζω ότι και ως πολιτικοί πραγματικά μπορούμε να μάθουμε πολλά από την ε, συμβολή σας αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι να συνεχίσετε με αυτή τη θέρμη, να εμπνέετε νέους ανθρώπους, να ε, παρακινήσετε και άλλους ε, ανθρώπους να βαδίσουν στα δικά σας χνάρια και πραγματικά με, με αγωνία περιμένω και το βραβείο της επόμενης χρονιάς. Θα ήθελα να πω ότι η νέα γενιά έχει κοινέ αξίες και όλοι θέλετε να συμμεριστείτε κοινέ αξίε και να μπορέσετε μέσω μουσικής ή μέσω αντιμετώπισης των προσφύγων να συνδράμετε σε αυτή την κοινωνία των νέων. Εγώ πολλές φορές έχω έρθει σε επαφή με νέους πρόσφυγες που έχουν γράψει βιβλία. Πρόκειται για ε, αυτοβιογραφίες που περιγράφουν τι έζησαν. Και αυτό για να υπάρχει μία πολιτισμική διαμεσολάβηση. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η προσωπική θεώρηση των πραγμάτων από τους πρόσφυγες. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς έχετε επαφή με τέτοιους εκδοτικούς οίκους. Εσείς ε, μέσω αυτών των δικτύων λαμβάνετε υπόψη κοινέ εμπειρίες. Υπάρχει και η Europa Canto στην Ιταλία, μια άλλη οργάνωση που ενώνει την Ευρώπη μέσω του τραγουδιού. Και ε, αναφέρεται ότι ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί παρά να γεννηθεί Ευρωπαίος. Αυτό είναι το, αυτή είναι η εμβληματική ρίση της οργάνωσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσατε να βρείτε και άλλες κοινέ αξίες και άλλα κοινά σημεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Helga Trüppel. Σας ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, τρεις προσκεκλημένους, δύο και μια κυρία. Ε, πραγματικά εμπνευσμένε οι ομιλίες σας. Είπε η Φαρά ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα να κλέψει τα όνειρά μου. Και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω σε 30 χρόνια που ασκώ την πολιτική και συχνά επιτυγχάνω αντιλαμβάνομαι γιατί αγαπάτε το Βερολίνο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βεβαίω και άλλε πόλει μου αρέσουν, αλλά το Βερολίνο είναι τόσο πολυπολιτισμικό και έχει συγκεντρώσει τόσου μετανάστε, ε, πρόσωπα από διάφορε άλλε χώρε, καλλιτέχνε, οι οποίοι ζουν και σε ένα ε, σημείο τομή ανάμεσα σε διάφορε υπήρου και ε, αυτό το μεγάλο χωνευτήρι έχει και ένα φίλο μου που είναι μια φίλη μου μάλλον, ε, ζει εκεί, είναι συγγραφέα εβραϊκής καταγωγής και λέει ότι της αρέσει περισσότερο εκεί από το Μανχάταν. Τώρα για την υπόθεση της όπερας. Να τίνετε το χέρι προς τους νέους, να τους κάνετε να κατανοήσουν γιατί η όπερα είναι τόσο θαυμάσια και προξαλεί τόσες συγκινήσεις και να δώσετε στις νέε και στους νέους να το καταλάβουν αυτό. Γιατί πολύ συχνά ακούω από αυτού που ασχολούνται με την όπερα ότι, να μου λένε ότι δεν φτάνουμε μέχρι του νέου. Αν μου επιτρέπετε θα το βάλω μάλιστα και στην ιστοσελίδα μου το σύνδεσμο. Και για εσά από την Πολωνία. Αν υπάρχει ευρωπαϊκή μνήμη. Η ερώτηση είναι πραγματικά σημαντική και πόσε φορέ την έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Ίσως να μην είναι μοναχα μια ενιαία ευρωπαϊκή μνήμη, αλλά ίσω να είναι συνδυασμό διαφόρων μνημών. Και συνολικά πρόκειται για μια σύνοψη μνημών, αν μπορεί να το πει έτσι. Σημασία λοιπόν έχει ότι δεν είναι μια και μοναδική, αλλά ένα πλήθος μνημών που όμως όλες εντάσσονται σε ένα ενίο σύνολο. Ίσως έτσι μπορούμε να διδαχτούμε εμένα από τους δε και να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα που έκαναν οι ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους αιώνες και τις τελευταίες δεκαετίες. Γι' αυτό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είστε εδώ και που κάνατε όλες αυτές, όλη αυτή τη θαυμάσια δουλειά και οι τρεις σας και παρακαλώ συνεχίστε. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος, η Julie Ward. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να μας μιλήσετε, για να μας κάνετε να νιώσουμε ελπίδα. Η ναι είναι η απάντηση για το μέλλον. Έχει μεγάλη σημασία το ότι βρίσκεστε εδώ και έχει μεγάλη σημασία αυτή η διαφοροποίηση προγραμμάτων. Εκπροσωπείται ε, μία ε, ευρεία πλευρά του ε, ακτιβισμού της Ευρωπαϊκής Νεολαίας μπορεί κανείς να εξερευνήσει, να διερευνήσει ιδέες, και να τις μεταδώσει σε άλλους. Εγώ είχα ασχοληθεί με τις θεμελιώδεις αξίες της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Οι 28 ε, υπουργοί παιδείας είχαν συνεδριάσει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δώσουν κοινέ απαντήσεις μέσα στα πλαίσια μιας διάσκεψης. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η επικοινωνία μεταξύ μας. Υπήρχε πολλής εθελοντισμός, συνάντηση ανθρώπων και ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που παρουσιάσατε και εσείς. Φάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ασχολούμαι στη χώρα μου με θέματα ΛΟΑΔ και βρέθηκα και στα Σκόπια το Σαββατοκύριακο γιατί εκεί έγινε μια εκδήλωση για την κοινότητα των ΛΟΑΔ. Ξέρω ότι γίνονται πολλές διακρίσεις εκεί και ιδιαίτερα οι τρανσεξουαλικοί αντιμετωπίζουν μεγάλο μίσος Κάνετε μία εξαιρετική εργασία, είσαστε μία ε, νέα γυναίκα που κάνει ό,τι μπορεί. Έχει σημασία το από πού προέρχεσαι, πώς επιβίωσες και τώρα έχεις ηγετικές ικανότητες. Είσαι ο αγγελιοφόρος ενός μηνύματος. Θα μιλήσω και στην κοινότητα των ε, ΛΟΑΔ για την δική σου ιστορία έτσι ώστε να διαδοθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους τρεις βραβευθέντες. Ακούστηκαν και κάποια ερωτήματα άλλωστε, τα οποία ίσως θέλετε να απαντήσετε. Ας ξεκινήσουμε από τη Φάρα. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα της κυρίας Κώστα. Ε, βρίσκομαι σε διαδικασία επαφής με κάποιους εκδότες. Η, το πρώτο μου βιβλίο ε, πουλήθηκε σε 18 αντίτυπα, 18.000 αντίτυπα, συγγνώμη, πήγε, πήγα σε σχολεία, μίλησα με νέους ανθρώπους, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία, μίλησα και με, ακόμη και με 10 παιδιά στην Νορβηγία, με 15χρονα παιδιά στη Φιλανδία, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν είχαν ε, αυτή την κακόβουλη, αν θέλετε, διάθεση, όπως είχαν κάποιοι ενήλικες που συνάντησα στο ταξίδι αυτό και αυτό νομίζω ότι αναδεικνύει και τη σημασία της, ε, της ε, κοινωνικής και διαπροσωπικής επαφής. Δυστυχώς όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι αρχίζουν ε, τα, τα, τα, αρνητικά. Το, η πρώτη γερμανική λέξη που έκφραση που έμαθα ήταν το «αχ, ζω». Α, έτσι λοιπόν. Και το ακούω αυτό πλέον κάθε μέρα και από τον φίλο μου, τον σύντροφο μου ε, ο οποίος κάθε μέρα ε, με υποδέχεται με αυτήν την ε, έκφραση του την, του την ανταποδίδω και εγώ. Είναι εξαιρετική πόλη πραγματικά η, το Βερολίνο. Το αχζό στα γερμανικά σημαίνει «Α, ωραία, κατάλαβα». Όταν σου λέει κάποιος κάτι μπορείς να πεις αχζό εννοώντας ότι «εντάξει, α, κατάλαβα». έγινε ε, ε, έδωσα και μια συνέντευξη κάποια στιγμή όταν δεν ήξερα ακόμα γερμανικά καθόλου και ε, μου απαντούσε ο δημοσιογράφος αυτή την έκφραση πάντοτε και γι' αυτό και μου προκάλεσε αυτή την εντύπωση και την απορία. Έμαθα όμως. Λοιπόν, το Βερολίνο είναι εξαιρετική πόλη, τα LGBT θέματα είναι πολύ σημαντικά για μένα. Δεν αντιμετωπίζω διακρίσεις ιδιαίτερες γιατί η η κοινωνία μας ε, είναι οπτική αν θέλετε. Στην κοινωνία μας, ε, στην, στην κοινότητα των LGBT, των διεμφυλικών συγκεκριμένα, το, το ε, ονομάζουμε αυτό passing. Δηλαδή με περνάνε για γυναίκα λόγω της εμφάνισής μου, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζω προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλοι, άλλα μέλη της κοινότητας LGBT. Ε, το Βερολίνο επίσης ήταν η πρώτη πόλη που συνέστησε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων από την ΛΟΑΔ κοινότητα. Αυτό επίσης ήταν εξαιρετικό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε σε άλλες χώρες οι πρόσφυγες ΛΟΑΔ απλά μπαίνουν στο, στα ίδια στρατόπεδα στους ίδιους καταβλισμούς με, κανονικούς, με straight πρόσφυγες και αυτό πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Και εγώ θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχήν σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας που μας τιμά. Ε, ως προς την όπερα στην Ευρώπη προσπαθούμε, προσπαθούμε να την διαδώσουμε. Δεν είναι όμως εύκολο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις και ίσως νέοι δεν είναι και άμεση προτεραιότητα γιατί εμείς δεν είμαστε μεγάλοι χρηματοδότες που συνδράμουμε ε, χρηματικά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άρα δημιουργούμε μία ε, σχέση με το θέατρο. Ο Βατσλάβης έλεγε ότι η σχέση βοηθάει και το περιεχόμενο. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει κανείς τι είναι το θέατρο, αλλά αν ένας φίλος του πει «Μα, έλα, θα δεις, θα περάσουμε καλά», τότε θα ζήσει αξέχαστες εμπειρίες. Μην ξεχνάμε την αρένα της Βερόνας. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει πείρα. Χρειάζεται να έχει ένα ζευγάρι αυτιά και καλή διάθεση. Δεν είναι εύκολο να ζητήσουμε ραντεβού με τον καλλιτεχνικό διευθυντή βεβαίως. Υπάρχουν διαμεσολαβητές που προσπαθούν όπως στο φεστιβάλ της Μάντοβας ε, προσπάθησε να μας βοηθήσει ναι. ο καλλιτεχνικός διευθυντής ε, Εμείς στη Γιουβενάλια προσπαθούμε να γίνει πιο προσπελάσιμη η όπερα στους νέους. Όταν ήμουνα ε, νέα ετών ζήτησα από τον πατέρα μου να με πάει στην αρένα της Βερόνας. Είδα την Αΐντα όπου γίνεται λόγος για διαφυλετική αγάπη. Ε, γίνεται λόγος ε, για τον πόλεμο επί δύο ώρες και η τελευταία λέξη είναι η ειρήνη. Ειρήνη, ειρήνη σε λατρεύω, λέει ο Αμνέρης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, ιδέες. Ας πούμε για παράδειγμα, κάθε φορά που πηγαίνω στο θέατρο ή στην όπερα, ε, νιώθω συγκλονισμένος. Είναι μεγάλες αυτές οι ιδέες. Τώρα, ως προς τους, την κοινότητα των ε, ΛΟΑΘ πρόκειται για μία κοινότητα που έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες. Δεν έχει σημασία η προέλευση. Υπάρχουν οι μεγάλες ορχήστρες ε, που διευθύνει, για παράδειγμα, ο Μπάρεμποιμ. Ε, έχουν περάσει 25 χρόνια από το θάνατο του Νουρέγευ που πέθανε από AIDS. Αλλά αν ακούσετε ε, μία άρια που είχε τραγουδήσει Μαρία Κάλλα στη σκάλα του Μιλάνο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλές ε, άριες τραγουδήθηκαν και από τραγουδιστές, τενόρους ή βαρύτονους οι οποίοι πέθαναν από AIDS. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τι είπε η δόκτωρ Τόμσον από την Ατλάντα που μίλησε για τους οροθετικούς και παρενέβη άμεσα και στον κόσμο του θεάτρου. Και πολλές φορές θεωρώ ότι τα λόγια από άριες της όπερας ε, λένε πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε διαφορετικά. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο Τόμας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, όλους και όλους που μιλήσατε. Ευχαριστώ επίσης τους οργανωτές ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι μοιράζονται την πίστη τους την πίστη τους στην ε, φύση του ανθρώπου. Ευχαριστώ επίσης αυτούς που ηγήθηκαν των καλλιτεχνικών εργαστηρίων. Είναι άνθρωποι που έχουν ασκήσει αυτή τη δραστηριότητα για ολόκληρη τη ζωή τους. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ήταν, μελετητές, ήταν φοιτητές της αρχιτεκτονικής, της αρχαιολογίας και άνθρωποι όπως εγώ. Που οι δικές μου σπουδές δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της συνάντησης αυτής. Η συνάντηση αυτή όμως είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συνάντηση ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικές χώρες. Είναι και συνάντηση ανθρώπων με πολύ διαφορετικά ενδιαφέροντα. Και γι' αυτό το λόγο επιθυμώ να ευχαριστήσω και πάλι τους οργανωτές. Πρόεδρο, σα Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και πάλι. Όλος ιδιαίτερος που ήρθατε σήμερα εδώ και παρουσιάσατε το έργο σας. Νομίζω ότι όσοι σας παρακολούθησαν έχουν εντυπωσιαστεί πραγματικά και το μόνο που μπορώ να πω είναι συνεχίστε την προσπάθεια, προσπαθήστε να εμπνεύσετε και άλλες νέες και νέους να παραγάγουν και άλλο νέο έργο. Συνεχίστε πάντως και με τα δικά σα αυτά που έχετε φτιάξει ω τώρα, τα οποία είναι πραγματικά θαυμάσια. Σα ευχαριστώ και πάλι. Και πολύ χαίρομαι που λάβατε, που βραβευθήκατε δηλαδή με το βραβείο Καρλου Α, τώρα θα, θα βγάλουμε και μια φωτογραφία. Αυτή τη λεγόμενη οικονομική, ε, με συγχωρείτε, οικογενειακή φωτογραφία. Δηλαδή τα εναπομένοντα μέλη τη Επιτροπή Πολιτισμού με του τρει βραβευθέντες, δηλαδή δύο και μία βραβευθήσα.